Ja, sehr Αγαπητοί κυρίε και κύριοι συνάδελφοι τη Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού, αγαπητοί προσκεκλημένοι, σα καλωσορίζω στην σημερινή μα συνεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι Βρυξέλλε. Έχουμε καταρχά να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Αν δεν έχετε αντίρρηση, την εγκρίνουμε όπω έχει υποβληθεί. Αντιρρήσεις δεν βλέπω. Α, όχι, η κυρία Τσέσκοβα έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, είδα στο πρόγραμμα ότι προβλέπετε να συζητηθεί δική μου έκθεση σήμερα και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρωτοβουλία να προβλέψετε το θέμα αυτό. διότι αρχικά είχε προβλεφθεί παράταση προθεσμιών μέχρι την έγκριση της ε, εκθέσεώς μου. Ερωτώ λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα για μια παράταση, για μια αναβολή καλύτερα για να ψηφίσουμε τον Ιούνιο, ώστε να έχουν και οι συνάδελφοι της Επιτροπής τη δυνατότητα να καταθέσουν τις τροπολογίες του. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Ο Πρόεδρος. Να ρωτήσω τη γραμματεία, ναι. Μάλιστα, είναι δυνατόν. Εάν συμφωνούν όλα τα μέλη της Επιτροπής, ευχαριστώ να δώσουμε την ε, παράταση. Και αν μου επιτρέπετε μια ακόμη λεπτομέρεια, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να είμαι βεβαία ότι θα γίνει ψηφοφορία όπως αρχικά είχε προβλεφθεί για την Ολομέλεια. Ότι δεν θα αλλάξει δηλαδή σε σχέση με την ψηφοφορία στην Ολομέλεια που προβλέπονταν αρχικά τον Ιούλιο. Έτσι. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε 17 Ιουνίου την ψηφοφορία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα. Μετά να δώσουμε προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Και μετά νομίζω ότι θα ήταν σωστό και έναντι των συναδέλφων της Επιτροπής να μην αλλάξει η ημερομηνία για την ψηφοφορία στην Σύνοδο του Ιουλίου, στις 10 Ιουλίου. ή μήπω πρέπει να περιμένουμε κάποια απάντηση από τον Πρόεδρο, δεν ξέρω. θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να αξιοποιήσω και τις, ε, τα αποτελέσματα των συζητήσεων από τις ακροάσεις. Γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα για την αναβολή αυτή, χωρίς όμως να σημαίνει ότι θα πρέπει και να καθυστερήσει μετά η ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Ε, ε, Ο πρόεδρο. Καλώς. Λοιπόν, το προβλέψαμε στην ευαρίστια διάταξη για σήμερα, αλλά πρέπει να σας πω ότι δεν είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να γίνει ψηφοφορία τον Ιούλιο, εάν η σημερινή συζήτηση αναβληθεί. Α το συζητήσουμε λοιπόν σήμερα όπως και να έχει, για να ξέρουμε ότι είμαστε σε θέση να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα και πολύ ευχαριστώ εντωμεταξύ θα επαληθεύσουμε εάν σε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας για την ψηφοφορία σε μπορεί πάντα να δηληθεί ε, το χρονοδιάγραμμα για ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Αλλά ας γίνει σήμερα η συζήτηση και αφήστε ένα περιθώριο να κοιτάξουμε. Εντάξει, συμφωνείτε. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Τσέσκοβα. Πολύ ωραία. Καλώς. Και άρα προχωρούμε με την ημερησία διάταξη. Επισημαίνω ότι έχουμε μετάδοση στο διαδίκτυο της εργασιών μας. Έχουμε τη διερμηνία, ως συνήθως. Και πρόκειται να γίνει η ηλεκτρονική ψηφοφορία μας. Θυμάστε ότι χρειάζεται να έχετε μέσα στην κάρτα σας όταν έρθει η ώρα για τις ηλεκτρονικές προφορές θα κάνουμε και μια δοκιμαστική βέβαια. Απλώς υπενθυμίζω ότι χρειάζεται η κάρτα και για την Τετάρτη. Και περνάω στο σημείο 3 με την έκρηση των πρακτικών της στις 18 18-19 Μαρτίου της τα πρακτικά αυτά δεν έχουν ε, δει ε, παρατηρήσεις ή ενστάσεις. Αν δεν έχετε εδώ αντιρρήσεις, μπορούμε να το εγκρίνουμε. Και προχωρώ στο σημείο 5 της ημερησίας διατάξεως, ορισμός μέλους του ελεκτικού συνεδρίου εκ μέρους της ε, κροατικής κυβερνήσεως προβάλλεται ως υποψήφιος ο κύριος Μάτεν, τον καλωσορίζω εδώ. Μάτες. Καλώς ήρθατε. Αρμόδια για την παρουσίαση της υποψηφιότητας είναι η κυρία Αιάλα Σέντερ. Με βάση το άρθρο 108 του κανονισμού πρόκειται να γίνει εδώ μία ακρόαση με τον υποψήφιο. Εν δε της ακροάσεως αυτής έχει δώσει απαντήσεις σε ένα ερωτηματολόγιο. Ο κάθε υποψήφιος έχει την δυνατότητα να κάνει μια εισαγωγική τοποθέτηση πεντάλεπτη και στη συνέχεια απαντά στις ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής και θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία εισηγήτρια να μας πει εάν έχει κάτι να συμπληρώσει η ίδια ή θα δώσω τον λόγο στον κύριο Νέβεν Μάτες για την εισαγωγική του παρατήρηση. Η κυρία Αγιάλα Σάντερα από ό,τι βλέπω δεν έχει αντίρρηση. Κύριε Μάτες, μια εισαγωγική παρατήρηση. Παρέμβαση παρακαλώ, πέντε λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας πω δύο λόγια για το πόσο σημαντική είναι αυτή η στιγμή για τους πολίτες της χώρας μου. Η Κροατία με την παράδοσή της, την ιστορία της, ανέκαθεν ανήκε στην ευρωπαϊκή οικογένεια των λαών και γι' αυτό ακριβώς ε, αυτή η στιγμή απέκτησε την πλήρη της ανεξαρτησία ε, δήλωσε υποψηφιότητα για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θεωρεί ότι εδώ συνενώνονται οι χώρες ε, για να αντιμετωπίσουν όλα τα θέματα της ε, ε, ζωής. Η διαδικασία προσχώρησης ήταν δύσκολη, η Κροατία προσπάθησε σκληρά να τηρήσει όλες τις προϋποθέσεις προσχώρησης και πλέον ο στόχος έχει επιτευχθεί. Γι' αυτό ακριβώς και χαιρόμαστε που οι προσπάθειές μας απέδωσαν καρπούς και είμαι περήφανος που είμαι ένα από του πρώτου κροατέ που προτείνεται για μία από αυτές τις τόσο σημαντικές θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα και ο πρώτος ο οποίος βρίσκεται ενώπιον ε, μιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ξεκίνησα την ε, καριέρα μου στο Ινστιτούτο Οικονομικών ε, του Ζάγκρεπ ως οικονομολόγος και τότε η χώρα είχε πολύ ψηλό πληθωρισμό και εγώ ασχολιόμουν ε, κυρίως με δημοσιονομικά ζητήματα και τη σχέση των, ε, της δημοσιονομικής κυριαρχίας ε, με την νομισματική πολιτική. Αργότερα ε, πήγα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όπως είπε και ένας από τους συναδέλφους μου, ένας από τους βασικούς ρόλους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου είναι κυρίως τα δημοσιονομικά ζητήματα. Ε, ασχολήθηκα με τα θέματα της βιωσιμότητας των ε, ε, δημοσιονομικών πολιτικών σε αρκετές χώρες και ασχολήθηκα και με προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής σε κάποιες χώρες και τις διάφορες δραστηριότητες του Ταμείου. Ασχολήθηκα και με διάφορα προγράμματα και αναπόσπαστο τμήμα της δημοσιονομικής πολιτικής ήταν να δούμε κατά πόσον η πολιτική που εφέρνουμε η χώρα ήταν βιώσιμη. Ένα από τα βασικά στοιχεία στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο είναι ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτά που έκανα ήταν επανομοιότυπα με αυτά που κάνει το Ελεγκτικό Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό ακριβώς και θεωρώ ότι ε, τα καθήκοντα που θα μου ε, αν και εφόσον μου ανατεθούν, θα είναι γι' αυτό το τομέα ιδανικά με ενδιαφέρουν θέματα ε, κατάλληλων λογιστικών ε, σε δημοσιονομικές διαδικασίες ε, και επίσης με ενδιαφέρει το ίδιο το θέμα των νομισματικών πολιτικών. Κυρίως τι γίνεται σε σχέση με την ε, ε κυβερνητική συνεργασία με μεγάλες επιχειρήσεις και ορισμένες φορές ε, βλέπουμε τι γίνεται με δημοσιονομικά θέματα διότι υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις που διεξάγουν δημοσιονομικά καθήκοντα αλλά εξαιρούνται από τον υπολογισμό τους ε, στη συνέχεια. Αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια κυρίως, όπως αποδείχθηκε και από την παρούσα κρίση, θα πρέπει ορισμένες φορές να δούμε τι κάνουν αυτές οι επιχειρήσεις, διότι ε, οι κυβερνήσεις αναγκάζονται να αναλάβουν το χρέος τους. Και φυσικά αυτό δεν βοηθά τις αγορές. Οι κυβερνήσεις βέβαια δεν είναι υπόψινες μόνο για τη συλλογή εσόδων και την εκτέλεση των προϋπολογισμών, αλλά συμμετέχουν και σε πολλές ε, οικονομικές διαδικασίες. Ε, από πλευράς ισοζυγίου πολλές φορές αναλαμβάνουν πολλές ευθύνες, και από πλευράς εσόδων το εξωτερικό χρέος χρειάζεται να υπάρχουν έσοδα για να μπορέσουν να καλύψουν ε, τις ε, εξωτερικές δαπάνες. Ορισμένε φορέ αυτέ οι δραστηριότητε θεωρούνται ότι βρίσκονται κάτω από τη γραμμή του προπολογισμού και δεν επηρεάζουν τον προπολογισμό ή δεν θεωρούνται σημαντικά στατιστικά στοιχεία ή αποκλείονται τελείω από του υπολογισμού του προπολογισμού. Υπάρχουν όμω ε, αφενό επιχειρήματα υπέρ αυτή τη διαδικασία, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρχει και πλήρη διαφάνεια σε αυτές τις διαδικασίες, διότι επηρεάζουν είτε άμεσα είτε όμεσα το δημόσιο χρέο. Ε, ο οικονομικός έλεγχος λοιπόν των δημοσίων λογιστικών δεν θα πρέπει να στέκεται απλώς και μόνον στην ακρίβεια των λογιστικών στοιχείων, αλλά θα πρέπει να αντιμετωπίζει και το θέμα των δημοσιονομικών κινδύνων, οι οποίοι απορρέουν από διάφορες κυβερνητικές δραστηριότητες που πολύ συχνά δεν περιλαμβάνονται στο γενικό προπολογισμό ενός κράτους. Αυτό είναι ένα θέμα βέβαια το οποίο απασχολεί περισσότερο τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή καθε αυτή. Αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση αναπτύσσεται και γίνεται ένας πιο περίπλοκος θεσμός και έχει και την προοπτική της Τραπεζικής Ένωσης, ο κίνδυνος αυτός γίνεται, λένε, και υψηλότερος και η σημασία του γίνεται πιο, πιο σημαντική. Ελπίζω λοιπόν ότι οι δεξιότητες που έχω αποκτήσει στο συγκεκριμένο τομέα θα μου επιτρέπουν να είμαι χρήσιμος για το ελεγκτικό συνέδριο όταν θα αναπτύξει και τις κατάλληλες δεξιότητες να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Με ενδιαφέρουν και θέματα δημοσίου χρέους σε μεγάλες οικονομίες. για κάποιο λόγο ακόμα πρέπει να τα εξηγήσουμε αυτά. Το δημόσιο χρέος έχει αλλάξει εδώ και 40 χρόνια και αυξάνεται συνεχώς ε, για κάθε χώρα. Συνήθως αυτό συμβαίνει σε καιρό πολέμου ή μεγάλης ύφεση, αλλά δεν συνέβη αυτό για τα τελευταία 40 ε, χρόνια. Ε, δυστυχώς ε, έχει μειωθεί σημαντικά ένας πολύ σημαντικός δημοσιονομικός χώρος, καθώς οι χώρες πλήττονται από την κρίση. Πολλές χώρες έχουν τεράστιες προκλήσεις για να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτά, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να διασφαλίσουν ότι θα μπορέσουν να έχουν και σαφή βελτίωση στα δημοσιονομικά τους. Το ελεγκτικό συνέδριο έχει στο θεματολόγιο του πολλά θέματα για το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δημιουργείται για να αντιμετωπίσει την παρούσα κρίση. Αυτό περιλαμβάνει και νέους μηχανισμούς για τη δημοσιονομική πειθαρχία και επίσης ε, και την πορεία προς τη Δημοσιονομική Ένωση. Όλα αυτά βέβαια προκειμένου να τεθούν σε εφαρμογή ε, σημαίνει ότι θα πρέπει και το ελεκτικό συνέδριο να τα ελέγχει και αυτός είναι σημαντικός ο ρόλος του. Επίσης διαπίστωσα ότι υπάρχει και μια σημαντική έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου για τη βελτίωση των στατιστικών στοιχείων για δημοσιονομικά ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ελέγχει επίσης και νέα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ε, και αυτό φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την έλεγχο και τη συμμόρφωση των ελέγχων δεν έχω και πολύ μεγάλη πείρα, αλλά ίσω θα μπορούσα να είμαι και μια φρέσκια ματιά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πολλά από τα έγγραφα του ελεγκτικού συνεδρίου με έκαναν να συνειδητοποιήσω ότι η έλλειψη συγκεκριμένων δημοσιονομικών πόρων δημιουργεί σημαντικέ προκλήσει. Υπάρχει ένα περίπλοκο ζήτημα εσωτερικών και εξωτερικών ελέγχων, πιστοποιήσεων και ελέγχων σε επίπεδο κρατών μελών, αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και ο τελικό πόλογο είναι φυσικά το ελεκτικό συνέδριο. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη χρήση των ευρωπαϊκών πόρων για να μπορέσουμε να έχουμε ομαλή λειτουργία αυτών των συστημάτων, ακόμα πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια πρόκληση. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι θα μπορούσαμε ίσως να εξετάσουμε το ενδεχόμενο να κινηθούμε προς μια κατεύθυνση που μας, μας επιτρέψει να συντονιστούμε καλύτερα για τη χάραξη πολιτική σε αυτή τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή βέβαια μόνο γενικές δηλώσεις μπορώ να κάνω, δεν μπορώ να είμαι πιο συγκεκριμένος, αλλά εάν με επιλέξετε για το ελεκτικό συνέδριο θα προσπαθήσω να είμαι πιο συγκεκριμένος. Ολοκληρώνοντα, κύριε Πρόεδρε, να σα πω ότι είμαι βέβαιο ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και οι δραστηριότητε του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι αλληλένδετα και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα από τα βασικά στοιχεία του ευρωπαϊκού συστήματος λογοδοσίας. Γι' αυτό ακριβώς δράτω με τις ευκαιρίες να σας πω ότι σε περίπτωση που επιλεγώ θα προσπαθήσω να συνεργαστώ όσο το δυνατόν καλύτερο με την Επιτροπή. Ε, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση εδώ στην ακρίωση και για το γεγονός ότι μου δώσετε τη δυνατότητα να σας ε, συστηθώ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάτες για την ε, εισαγωγική σας παρέμβαση. Να δώσω τώρα το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Η γήτρια καταρχάς, η κυρία Ινέσα Γιάλα Σέντερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κύριε Μάτες στην ακρόαση. Διάβασα πολύ προσεκτικά όλες τις ε, απαντήσεις που δώσατε και διάβασα και κάποια άρθρα τα οποία έχετε συγγράψει για την κατάσταση στην Ελλάδα. Ένα άρθρο το οποίο με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι ε, στάθηκε πολύ στα σφάλματα, κάτι το οποίο... Ε, συνήθως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την τάση να λησμονούμε και πολλές φορές επαναλαμβάνουμε και τα ίδια λάθη του παρελθόντος. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να το επισημάνετε αυτό και θεωρώ ότι είστε κάποιος ο οποίος εκπείρας είναι σε θέση να αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν και θέλει να μάθει από τα λάθη. Από το βιογραφικό σας σημείωμα βλέπουμε, και το είπατε κι εσείς, ότι δεν γνωρίζετε πολλά πράγματα όσον αφορά τα θέματα συμμόρφωσης. Ε, έχετε βέβαια μια εντυπωσιακή σταδιοδρομία, δεν είστε απλός και μόνο ένας οικονομολόγος, γνωρίζετε πάρα πολλά πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν αφορά τα νέα μέσα για την ε, ε, Τραποζική Ένωση και τη Δημοσιονομική Ένωση, τα οποία δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία συζητούν αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται μία απόπειρα να ελεγχθούν αυτά τα μέσα. Αυτό προσπαθεί να κάνει και το Κοινοβούλιο αλλά και το Ελεγκτικό Συνέδριο. Εσείς Πώς θεωρείτε ότι μπορεί να βοηθήσει η πείρα σας όταν θα πρέπει να βρείτε τρόπους μέσω των οποίων το ελεκτικό συνέδριο θα μπορεί να ελέγξει πιο αποτελεσματικά όλα αυτά τα νέα μέσα δανειοδότησης εγγυήσεων τα οποία δημιουργούμε αυτή τη στιγμή και δημιουργούν και μία δομή κάπως περίπλοκη και περίεργη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι ακριβώς θεωρείτε ότι χρειαζόμαστε, διότι αυτή τη στιγμή ε, τι έχουμε. Ένα μέλος του ελεκτικού Συνέδριο που συμμετέχει μεν, αλλά το ελεκτικό συνέδριο αυτό καθεαυτό κατά την άποψή μας δεν είναι απόλυτα ενταγμένο σε αυτή τη διαδικασία ελέγχου των νέων μέσων και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε λίγο περιορισμένη και δεν μπορούμε να ελέγξουμε όσο θα θέλαμε. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. digamos, eh, distinta, distinta τα έχετε πείρα για τα προγράμματα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γνωρίζετε, φαντάζομαι κι εσείς, ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή να εξελίξει μια συζήτηση ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση τους τελευταίους μήνες και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πώς μπορούμε να ε, συμφιλιώσουμε τα προγράμματα λιτότητας έχοντας συνεχώς και κατά νου την ανάγκη να υπάρχει μια ισορροπία με προγράμματα επενδύσεων και ανάπτυξης. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε αν μπορείτε εσείς ε, από την πείρα σας να μας βοηθήσετε και να μας πείτε και την άποψή σας για το θέμα αυτό. Και τέλος, στο βιογραφικό σας σημείωμα έχει κάτι το οποίο μου δημιουργεί ένα ερώτημα. Είστε στο ε, Προεδρείο, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Οικονομικών του Ζάγκρεπ. Θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς κάνετε σε αυτό το Ινστιτούτο. Μια τελευταία ερώτηση, την οποία κάνουμε σε όλους τους υποψηφίους ε, για μέλη του ελεκτικού συνεδρίου. Είστε διατεθειμένος να παραιτηθείτε από αυτή τη θέση σε περίπτωση που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχει αντίθετη άποψη ε, Μας δίνετε μια ευφυή απάντηση, αλλά εγώ δεν ξέρω τι επαρκεί. Εάν το Κοινοβούλιο αποφασίσει ε, κατά της υποψηφιότητάς σας, εσείς τι θα κάνετε. Yeah, thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Μάτες. Ευχαριστώ. Και ας ξεκινήσω από το εύκολο, το οικονομικό του Ζάγκρεπ. Το 1992 εργάστηκα εκεί, μετά ανέλαβα καθήκοντα σε διάφορε θέσει, δεν ξέρω αν θα τι θυμηθώ όλε. Πρόσφατα πάντως ήμουν πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχει όμως εκπνεύσει πλέον η θητεία μου. Δεν είμαι πλέον δηλαδή πρόεδρος ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο. Λιτότητα και ανάκαμψη ναι, όθηση στι ευρωπαϊκέ οικονομίε με προβλήματα. Βέβαια η ανταγωνιστικότητα θα είναι το πρώτο και κύριο. Σε έναν βαθμό μπορούμε πιστεύω να αξιοποιήσουμε τι επιτυχείς εμπειρίες μια χώρα που δεν είναι χώρα τη Ευρωζώνης, αλλά ε, δρούσε σε ένα περιβάλλον σταθερή ισοτιμία στη Λετωνία και η οποία επέτυχε να βγει από την δύσκολη κατάσταση συνδυάζοντας ε, μεταρρυθμίσεις αρκετά δύσκολες, αρκετά σκληρές. Βέβαια δεν πρέπει να λησμονούμε ότι κατά την ίδια περίοδο υποφελήθηκε από πολύ σημαντικά κονδύλια από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η καθαρή μεταφορά κονδυλίων για την περίοδο αυτή, δηλαδή της προσαρμογής, ήταν τεράστια. Άρα, και σκληρές μεταρρυθμίσεις, αλλά και χωρίς να θέλω να αναφέρω διεξοδικά ένα ολόκληρο κατάλογο ε, μέτρων, αλλά πάντως ήταν πάρα πολύ σκληρά τα μέτρα λιτότητας σε σχέση με αυτά που είδαμε σε άλλες χώρες, μαζί με σημαντική ενίσχυση μεταφορές κονδυλίων καθαρές και νομίζω ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει μια ε, θετική εμπειρία. Επίσης, Μια άλλη χώρα η οποία δεν αντιμετώπισε κρίση, αλλά πάντως μπήκε σε, αυτήν την, σε αυτούς τους κλειδονισμούς παγκόσμιους, όπως η Πολωνία, και που επίσης υποφελήθηκε από καθαρές ε, μεταφορές κονδυλίων. Και τα δύο νομίζω πρέπει να συμβαίνουν. Συνδυασμό δηλαδή σκληρών μεταρρυθμίσεων και στήριξη, για να το πω έτσι. Επίσης δεν θέλω να φερθώ στα νέα θεσμικά όργανα που θεσπίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη. Ναι, υπάρχει ο χαρακτήρας των διακυβερνητικών συμφωνιών για τα όργανα αυτά συνεπάγεται μια ιδιάζουσα δομή, λειτουργία που καθιστά πιο δύσκολη και την παρέμβαση του ελεκτικού συνεδρίου. Από την άλλη μπορούν ίσως να επιτελέσουν πιο ευχερό το έργο της επαλήθευσης των όσων συμβαίνει στη χώρα εκ μέρους του ελεγκτικού συνεδρίου. Με το ευρωπαϊκό εξάμεινο και το six-pack. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να συμβάλλει οπωσδήποτε το ελεγκτικό συνέδριο στην παρακολούθηση μέσω του ελέγχου των πρόοδων στις, ε, στους τομείς αυτούς, κατά πόσο είναι συνεπής η προόδος στις διάφορες χώρες, χώρες τι επιτυγχάνεται. Αυτά. Σε αυτό το σημείο. Ε, επίσης, με καλύτερα να ε, επανατοποθετηθώ ή να επαναλάβω καλύτερα την απάντηση στη δεύτερη ερώτηση, στην τελευταία ερώτηση. Κοιτάξτε, οι κανόνες είναι ξεκάθαροι. Δεν διεκδικώ εγώ την ε, ικανότητα να αλλάξω κανόνες. Αλλά θα σας το πω ανοιχτά ότι αν τυχόν δεν έχω την υποστήριξή σας, κατά πάσα πιθανότητα θα αποσυρθώ. Να σας πω ότι εν πάση περιπτώσει εγώ θα αποσυρθώ, ή αν δεν με ότι οπωσδήποτε θα αποσυρθώ, θα συνεπαγόταν ε, εκ μέρους μου παραβίαση των αλλαγή των κανόνων. Θα έλεγα λοιπόν, το μόνο που μπορώ να πω σε αυτό το στάδιο είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα θα αποσύρω την υποψηφιότητά μου. Ευχαριστώ. Κύριος Οντή, παρακαλώ, εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο. Euh, je vous souhaite la bienvenue, euh, cher monsieur, et je voudrais dans le prolongement euh, ma collègue, je voulais vous poser la même question d'ailleurs. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας πω ότι λυπούμε για την απάντηση που δώσατε στην ερώτηση. Παρόλο που δώσατε μία γραπτή απάντηση, τη διάβασα, παρόλα αυτά θεωρώ ότι μετά την ψηφοφορία, όπως ξέρετε, εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τον υποψήφιο και συνήθως, συνήθως αποσύρεται η υποψηφιότητα μετά την ψηφοφορία. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η δική σας θέση αυτό, εγώ το σημειώνω. Έχετε μια εξαιρετική, αν θέλετε, υποψηφιότητα. Η υποψηφιότητα αυτή της Κροατίας είναι πραγματικά εξαιρετικά καλή και αν η εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου σας δοθεί, βεβαίως θα ακολουθήσει η αξιολόγηση. Το θέμα της αξιολόγησης των δημόσιων πολιτικών, όπως ξέρετε, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την απαλλαγή, αλλά είναι και το λεγόμενο αδύναμο σημείο της. Η Επιτροπή έχει καταλάβει αυτή τη διαδικασία βεβαίως, όπως και εμείς, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς θα μπορούσατε να συνεισφέρετε όσον αφορά τον έλεγχο των αξιολογήσεων βάσει των οποίων εμείς το Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να ε, ελέγξουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλος, συμπληρωματική ερώτηση, όσον αφορά το audit. Δεν έχετε ιδιαίτερη εμπειρία στον ε, έλεγχο. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, ρωτήσω αν ε, συμμετάσχετε τελικά στο ελεγκτικό συνέδριο. Φυσικά η η δήλωση, η δήλωση αξιοπιστίας που θα γίνει βάση του ελέγχου που θα κάνει το συνέδριο και βασίζεται στους διεθνείς λογιστικούς κανόνες, αυτούς που διέπουν κάθε τέτοιου είδους έλεγχο, είναι κάτι που είναι δεδομένο. Εσείς που δεν έχετε ιδιαίτερη εμπειρία στα θέματα αυτά, ιδιαίτερα στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, προτίθεστε να κάνετε κάποια ειδική κατάρτιση για να ενημερωθείτε καλύτερα με τα θέματα αυτά. Σας ευχαριστώ. Κοιτάξτε, όντως ε, ο τομέας αυτός δεν είναι ένα τομέα στον οποίο έχω ιδιαίτερη εμπειρία. Έχω όμω ε, μελετήσει όλε τι εκθέσει ε, του ελεγκτικού συνεδρίου και πολλέ ε, φορέ είδα ότι υπάρχουν σφάλματα όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, του κοινοτικού προϋπολογισμού, που εντοπίζονται από το ελεγκτικό συνέδριο. Ναι, εγώ μπορώ να παρακολουθήσω μια τέτοια διαδικασία. Ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις ε, δυσκολίες δεν είναι εύκολο να επιληθούν, κάποιες ναι. Για κάποιες ε, περιπτώσεις δεν έχω να προτείνω κάτι. Όσον αφορά την ε, συμμόρφωση Βεβαίως και είναι πολύ σημαντικές αυτές οι επιμέρους διαδικασίες γιατί τελικά με αυτόν τον τρόπο δίνεται και η τελική απαλλαγή και εγκρίνεται ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, όσον αφορά τις ε, δικές μου δεξιότητες και δυνατότητες να συνεισφέρω. ας πούμε ότι έχω σε κάποιους ε, τομείς λιγότερες ε, λιγότερη εμπειρία και λιγότερες, ε, ειδικο, λιγότερη ειδικότητα. Αλλά νομίζω ότι μπορώ να ανταπεξέλθω στο έργο εάν διοριστώ και επιλεγώ στο ελεκτικό συνέδριο. Ευχαριστώ πολύ, ο Γιάννη Πίλτερ. Γιάννη ε, Μόλτερ. Καλώς ορίσατε στην ε, Επιτροπή Ελέγχου του Προπολισμού. Είστε ο πρώτος εκπρόσωπος ενός νέου μέλους. Έχω μια γενική και μια ειδική ερώτηση να σας κάνω. Η γενική είναι ότι σκοπός και έργο του Ελεκτικού Συνεδρίου είναι να γνωμοδοτήσει όσον αφορά τους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως υπάρχει ένα ποσοστό σφαλμάτων της τάξης του 2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και 18 χρόνια και έχουμε ξεπεράσει κάθε φορά αυτό το ποσοστό 3,7 ήταν την τελευταία φορά και πολύ περισσότερο, παραδείγματος χάρη, για τα περιφερειακά ταμεία. Έχετε κάποιες προτάσεις για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και πώς συγκρίνετε την κατάσταση με την κατάσταση που ισχύει στην χώρα σας, στην Κροατία. Ποιο είναι το ποσοστό σφαλμάτων. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη πιο ειδική. Δεν ικανοποιήθηκα με την απάντηση που δώσατε. Σε περίπτωση που η γνώμη της Επιτροπής μας είναι αρνητική. Αν είναι αρνητική, σκεφτείτε το. Πώς, αν τελικά αποφασίσετε να παραμείνετε, θα συνεργαστείτε με μια επιτροπή που δεν σας έχει εκβάσει την εμπιστοσύνη της. Θα ξεκινήσω με την ειδική ερώτηση. Νομίζω ότι Όπως είπα, είναι μια περίπτωση η οποία δεν νομίζω ότι θα συμβεί. Κοιτάξτε, έγραψα αυτό που έγραψα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μακρηγορήσουμε για το θέμα αυτό. Φυσικά και θα λάβω πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μου την γνωμοδότηση και πιθανότατα θα αποσυρθώ. Αλλά βεβαίως θα ζητήσω να μου αιτιολογήσετε αυτήν την απόρριψη. Και βεβαίως σε αντίθετη περίπτωση, αν υπάρχουν όντως αντιρρήσεις, πιθανότατα θα αποσυρθώ. Τώρα, στην γενική σας ερώτηση, ναι, όντως και μένα με εντυπωσίασε η συχνότητα των ε, σφαλμάτων, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν ε, πολλές περιπτώσεις που μπορεί να συμβαίνουν εδώ. Παραδείγματο χάρη, εάν επαναλαμβάνονται τα σφάλματα, ίσως αυτό οφείλεται στο ότι δεν έγιναν οι επαιτούμενες ε, διορθώσεις, διευθετήσεις. Εάν η κάθε χώρα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες στο έπακρο, αν αυτή είναι, αν θέλετε, η στάση και των ε, οργάνων ελέγχου και εποπτείας επιτήρησης, και κοιτώντας το ιστορικό του επίπεδου των σφαλμάτων που υπάρχουν, πιστεύω ότι κάτι θα έπρεπε να γίνει. Εν πάση περιπτώσει, δεν θα σας κάνω προτάσεις εδώ, σε αυτό το στάδιο που βρίσκομαι. Ίσως σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις σφαλμάτων, θα μπορούσε να μειωθεί η, διαχείριση, επιμερισμένη διαχείριση. Ή θα μπορούσε κανείς να φανταστεί έναν μηχανισμό όσον αφορά την χρήση αυτού του 100% ή ενός πολύ μεγάλου ποσοστού των διαθέσιμων πόρων. Και αναρωτιέμαι γιατί το ονομάζουμε δήλωση. Ενδεχομένως θα έπρεπε, θα ήταν πιο σωστός τίτλος, να ονομαζόταν εθνική έκθεση, έκθεση των κρατών αυτή. Λέγοντας ότι αυτό είναι το ποσό που χρησιμοποιήθηκε. Και σε αυτή την περίπτωση να δίνεται και μια τεκμηρίωση όσον αφορά τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν αυτά τα κονδύλια, αυτοί οι πόροι. Ξέρω ότι κάποιες χώρες το κάνουν με έναν πιο επίσημο τρόπο. Δεν ξέρω, ίσως αυτές οι εθνικές εκθέσεις θα έπρεπε να παρουσιάζονται με ένα πιο τεκμηριωμένο και ολοκληρωμένο τρόπο όσον αφορά την χρήση των κονδυλίων. Αυτά. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω στο στάδιο που βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάτες. Δεν έχουμε άλλες ερωτήσεις. Α, μία μικρή ερώτηση. Σας ευχαριστώ, κύριε Σοντή. Μία διευκρίνηση, για να είμαστε σαφείς. Οι δύο συνάδελφοι αναφέρθηκαν στην απόφαση του υποψηφίου μετά από αρνητική γνωμοδότηση. Δεν αναφερόμασταν στην γνωμοδότηση εδώ της Επιτροπής μας, αλλά του Κοινοβουλίου. Αναφερθήκατε στην Επιτροπή, εδώ, σε αυτή την Επιτροπή. Η ερώτηση όμως που σας κάναμε είναι, θα αποσύρετε την υποψηφιότητά σας αν είναι αρνητική στάση του Κοινοβουλίου. Πρόεδρος, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί εμείς εδώ απλώς εκθέτουμε την ε, δική μας ε, σύσταση, την υποβάλλουμε, το κοινοβούλιο αποφασίζει. Ο κύριος Άντεργκαρδό όμως έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στην Επιτροπή. Έχω κι εγώ μία ερώτηση που αφορά μια πρόσφατη έρευνα που δείχνει ότι η διαφορά στην Κροατία είναι εξαιρετικά σημαντική. Είναι μία από τις πιο διαθαλμένες χώρες στην Ευρώπη. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Έχετε κάποιες προτάσεις, κάποιες σκέψεις. Πώς ε, μπορείτε να εξηγήσετε αυτή την ε, διαπίστωση. Και αυτή η διαφορά πώς επηρεάζει τις σχέσεις που έχει η χώρα σας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να μου απαντήσετε, θα ήθελα να ακούσω από σας πώς βλέπετε το θέμα της διαφθοράς στη χώρα σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ και εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση πολύ σύντομα. Πώς βλέπετε το θέμα της εφαρμογής ε, των ε, μέσων στην Κροατία. Ξέρουμε πολύ καλά τι είναι οι σχέσεις της κυβέρνησής σας ε, με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Θα αναφερθώ και στο ίδιο που σας προανέφερε ο συνάδελφος Σόντεργατ, το Ελεκτικό συνέδριο έχει άμεσες σχέσεις με τις ε, χώρες μέλη και ξέρω ότι υπάρχουν πολλές φορές προσπάθειες κάποιου μέλους μιας χώρας να καλύψει κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν η χώρα του. Πώς θα αντιμετωπίζετε εσείς ε, αυτό το θέμα, Πρόεδρος. Κύριε Μάτις, θέλετε να απαντήσετε σε αυτές τις τρεις τελευταίες ερωτήσεις. Ε, ξέχασα έναν συνάδελφο, κύριε Νάζο. Όχι, πρόεδρε, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις, θα ήθελα να ρωτήσω, ο κύριος Έρενχάουζερ, είσαστε κατά των εθνικών δηλώσεων αξιοπιστίες και των υποχρεωτικών αυτών δηλώσεων. Μπορείτε να μας κάνετε μια ευκρίνηση για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Ε, μιλάτε για το management declaration τότε, έτσι, μάλιστα. Να μας απαντήσει ο κύριος Μάτες. Μια σειρά από ερωτήσεις περιμένουν. για τη διαφθορά καταρχάς και τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την ε, προετοιμασία για την προσχώρηση, η Κροατία συνεργάστηκε στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ετοιμάσει μια σειρά από ε, διαδικασίες, έχουν προχωρήσει διαδικασίες ανακριτικές για την πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτό αφορά όχι μόνο τον Πρωθυπουργό, αλλά και τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό, Υπουργό Άμυνας, Υπουργό Γεωργίας. Άρα πιστεύω ότι αποδεικνύεται, όσο τουλάχιστον μπορεί κανείς να περιμένει από τις ανακριτικές αρχές, ότι έχει αναλυφθεί δράση. Αυτό μπορώ να δώσω ως απάντηση στην ερώτησή σας. Για τη διάκριση τώρα. Κοιτάξτε, δεν φαντάζομαι μεταξύ, Ευρωπαϊκής, ε, μεταξύ Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και Κοιτάξτε, εγώ δεν φαντάζομαι, να το πω ξεκάθαρα, ότι μπορώ να έρθω αντιμέτωπο με το κοινοβούλιο. Εάν το κοινοβούλιο δεν με ψηφίσει, αποσύρω την ε, ψηφιότητά μου. Να το πω ξεκάθαρα. Το Εθνική δήλωση είπα ότι με προβληματίζει ο όρος δήλωση. Νομίζω ότι έκθεση θα ήταν πιο σαφής όρος και θα εξηγούσε μια γενική υποχρέωση των εθνικών αρχών να λογοδοτήσουν για τον τρόπο με τον οποίο αξιοποίησαν ευρωπαϊκά κονδύλια. Έχω κάθε σεβασμό και υποστηρίζω πλήρως τον ε, μηχανισμό αυτόν. Από ό,τι βλέπω υπάρχει σημαντική απόκληση μεταξύ των όσων συμβαίνουν κάποια, από κάποιες πλευρές των κυβερνήσεων, από κάποια τμήματα και των όσων ε, κάνουν κάποια άλλα ε, υπουργεία. Αυτό λοιπόν. Είναι ένα γενικότερο ζήτημα, το ζήτημα της αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων. Μια γενικότερη λοιπόν εθνική έκθεση για το πώς αξιοποιήθηκαν οι πόροι θα ήταν για μένα η σωστή, η σωστότερη διατύπωση. Ε, πώς έχω λησμονήσει κάτι μιλή, καλύψαμε το θέμα της, ε, των δηλώσεων διαχείρισης. Τίποτα άλλο για, τα, για τους βουλευτές. Όχι. Ευχαριστούμε κύριε Μάτες. Ωστόσο, δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για να κλείσει. Παρακαλώ. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω απλώς τον κύριο Μάτες, ο οποίος ε, τελικώς διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν σας υποστήριξει, είστε διατεθειμένοι να αποσύρετε την υποψηφιότητά σας. Ε, αυτή εκλαμβάνω ως απάντησή σας. Θα ήθελα όμως ε, να σας πω ότι πραγματικά με ένα προφίλ σαν το δικό σας και επειδή εμείς θα θέλαμε πραγματικά να υπάρχει κάποια μορφή ελέγχου για αυτά τα νέα μέσα τα οποία δημιουργούνται, παρά το γεγονός ότι έχετε και εσείς δίκιο ότι ε, σε διακυβερνητικό επίπεδο υπάρχουν ίσως και περισσότερες δυσκολίες, αλλά σίγουρα χρειάζεται και μια κάποια δημιουργικότητα από πλευρά μελών του ελεγκτικού συνεδρίου, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει τη δυνατότητα δημοκρατικού ελέγχου για τα όσα γίνονται ε, και το πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέσα και με ποιο τρόπο θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά με την πείρα σας λοιπόν και την πείρα που έχετε στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο και τις σχέσεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κοινέ αποστολής ε, και ούτω καθεξής, θα ήθελα απλώς να σας ρωτήσω για να ολοκληρώσουμε αν ε, θα ήσασταν διατεθειμένος σε περίπτωση που ε, αναλάβετε καθήκοντα ως μέλος του, του Ελεγκτικού Συνεδρίου ε, να συνεργαστείτε με την Επιτροπή Ελέγχου του προπολογισμού, για να μπορέσουμε να έχουμε και αυτές τις δραστηριότητες που θα θέλαμε να διεξάγει το ελεγκτικό συνέδριο ώστε να γίνεται ένας αποτελεσματικός δημοκρατικός έλεγχος των μέσων για την ε, δημοσιονομική και οικονομική διακυβέρνηση που δημιουργούνται τώρα και που, για τους οποίους ε, οι πολίτες συχνά έχουν ερωτηματικά. Oh, thank you very Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάτες, σαφώς ούτως ή άλλως το ελεγκτικό συνέδριο γνωμοδοτεί και κάνει προτάσεις. Δεν είναι αυτό το οποίο αποφασίζει. Ε, επομένως, ο μόνος τρόπος να είναι αποτελεσματικό το ελεγκτικό συνέδριο είναι να συνεργάζεται με αγαστό τρόπο με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σας. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη η στενή συνεργασία, ιδίω στα θέματα στα οποία σταθήκατε εσεί, ε, διότι αυτό το θεσμικό πλαίσιο είναι υπό ανάπτυξη. Ε, δεν έχει ακόμα καθοριστεί ούτε η διαδικασία, θα είναι κάτι το περίπλοκο. Δεν υπάρχουν λοιπόν εύκολες λύσεις, αλλά όπως είπατε και εσείς υπάρχουν και κάποια νομικά ε, προβλήματα τα οποία σχετίζονται με τα μέσα αυτά. Θεωρώ λοιπόν ότι συντρέχουν οι λέγοι για ε, στενή συνεργασία και δεν νομίζω ότι θα έπρεπε κάποιος να μη συνεργάζεται. Σας ευχαριστώ. Απαντήστε στις ερωτήσεις μας. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού προφανώς θα το αντιλαμβάνεστε. Θεωρεί ότι έχει κέρια σημασία συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό άλλο το καταγράφουμε παγίως και στη σχέση μας με την Όλαφ. Σας ευχαριστώ κύριε Μάτες. Uh-huh. we to... little uh, Θα κάνουμε τώρα ένα σύντομο διάλειμμα. Πολύ σύντομο. Και προσκαλούμε τώρα τον υποψήφιο που έχει υποστηρίξει η κυβέρνηση της Ρουμανίας. Παρακαλώ. Ο κύριος Πούφαν. Ja, liebe Mitglieder des Ausschusses für Haushaltskontrolle, ich darf in der Tagesordnung direkt äh, fortfahren. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού, έχουμε τον δεύτερο υποψήφιο για την θέση του Διευθυντού του Ελεκτικού Συνεδρίου μας έχει προταθεί από την κυβέρνηση της Ρουμανίας. Είναι ο κύριος Πούφαν. Δεν ξέρω αν προφέρω σωστά το όνομά σας. Κύριε Πούφαν, δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε υποψήφιο να πάρει το λόγο για πέντε λεπτά. Μας έχετε ήδη απαντήσει βάσει του ερωτηματολογίου. Σας έχουμε στείλει ένα ερωτηματολόγιο. Κατόπιν τα μέλη της Επιτροπής έχουν τη δυνατότητα να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Και βεβαίως ε, θα δώσω το λόγο πρώτα στην εισηγήτρια. Κύριε Πούφαν, έχετε το λόγο όμως καταρχήν για λίγα λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ, ενώπιόν σας. Ο διάλογος αυτός με τιμά. Ύστερα από την ακρόαση. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να ξαναέρθω, να προχωρήσω μια ευάθυνση στην ανταλλαγή απόψεων και διάλογο στα θέματα κύριου ενδιαφέροντος, όπως έχουν περιγραφεί, και που έχουν βέβαια, όπως συμφωνούμε όλοι, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον Ευρωπαίο πολίτη. Και τώρα με την αδειά σας, θα ήθελα εν συντομία να σας ε, παρουσιάσω κάποια στοιχεία της επαγγελματική μου δραστηριότητες και ελπίζω στη συνέχεια να απαντήσω ικανοποιητικά στα ερωτήματα που μου απευθύνατε επαγγελματική μου διαδρομία περιστρέφεται γύρω από το Ρουμανικό Ελεγκτικό Συνέδριο όπου ξεκίνησε το Μάιο του 1994 περνώντας τον διαγωνισμό για εισαγωγικές εξετάσεις στο σώμα των δημοσίων υπαλλήλων και είμαι ύστερα από άλλο διαγωνισμό ε, 20 χρόνια αργότερα, Γενικός Γραμματέας, κύριος Διατάκτης. Αυτό έχει και βέβαια επαγγελματική, επαγγελματικό κύρος, αλλά και ηθικό κύρος μεγάλο. Είχα σε όλη αυτή τη διαδικασία περίπλοκια καθήκοντα όπως τον συντονισμό των εφιστομενών διευθύνσεων, των περιφερειακών λεκτικών τμήματων και πέραν της ε, διαχειριστικής ικανότητας και δεξιότητας απαιτούνταν και ικανότητες συντονισμού και ικανότητες λήψη αποφάσεων μερικές φορές δύσκολων, ιδιαίτερα σε περιόδους δημοσιονομικής λιτότητας, περιορισμό δηλαδή των δαπανών και ορισμό προτεραιοτήτων. Πέραν της επαλήθευσης της διαχείρισης των πιστώσεων, με την οποία είναι επιφορτισμένο το Λεπτικό συνέδριο, είχα και τον έλεγχο της αποτελεσματικής χρήσης των κονδυλίων, όπως ορίζει ο νόμος, και την παρουσίαση των λογαριασμών, το συντονισμό του λογιστικού έργου, και την παρουσίαση ενώπιον της Βουλής των, της κάτω και της άνω βουνής, της Βουλής και της Γερουσίας δηλαδή, και των αρμοδίων επιτροπών, των σχετικών λογαριασμών από το ελεγκτικό συνέδριο. Το ελεγκτικό συνέδριο της Ρουμανίας, ε, πέραν του ελεγκτικού του έργου, καταρτίζει και παρουσιάζει και το δικό του προπολογισμό, ο οποίος υφίσταται τη διαδικασία έγκρισης από τα κοινοβουλία, από τις βουλές. Πρόκειται για μια αρμοδιότητα βεβαίως που ανήκει στο Γενικό Γραμματέα, υπήρχε όμως στην, ε, στο συντονισμένο όργανο των δύο βουλών, της Κάτω και Άνω της Ρουμανίας, ο έλεγχος του προπολογισμού αυτού και ποτέ δεν βρέθηκε, ποτέ δεν καταγράφηκε κάποιο αρνητικό αποτέλεσμα. Έχω επίσης αναλάβει το συντονισμό των προγραμμάτων υποστήριξη ε, των εξωτερικών προγραμμάτων που είχε αναλάβει το ηλεκτρικό συνέδριο για την ανάπτυξη και θέσπιση ελέγχου των λογιστικών με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και βέβαια αντίστοιχες δυνατότητες κατάρτισης προκειμένου να τηρήσουμε αυτές, να τηρήσω αυτές τις προδιαγραφές, προχώρησα στην βελτίωση, οργάνωση, μεθοδολογική προσέγγιση, προσδιορισμό κριτηρίων, προκειμένου να προσδιοριστεί ένα σύστημα δημοσιονομικού ελέγχου, προσδιορίσε ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου με τα μέτρα που το συνοδεύουν και ως κύριος διατάκτης των πιστώσεων είχα την αρμοδιότητα της καθοδήγησης των ειδικών δραστηριοτήτων για την ε, χορήγηση εντολής, εκτέλεση και εκαθάριση λογαριασμών για το κράτος. Το 2003 ήμουν μέλος μιας ομάδας θεσμικής, ε, θεσμικού χαρακτήρα για την υπαγωγή του ελεγκτικού συνεδρίου με βάση την ε, νομοθεσία που εξεργαστήκαμε στην δικαιοδοσία των αρμοδίων δικαστηρίων. Έτσι λοιπόν αναδιοργανώσαμε στην περίοδο που ήμουν εγώ στο Ελεκτικό Συνέδριο τις, ε, τα δημόσια οικονομικά, τη λειτουργία του Ελεκτικού Συνέδριου. Και σημειώνει μεγάλες αλλαγές στο Ελεκτικό Συνέδριο με βάση και τις αρχές της λειτουργίας του, την απλούστευση και την εκτέλευση των λογαριασμών. Με την ουσιαστική αυτή αλλαγή με την επαλήθευση εκ των υστέρων. Το ελεγκτικό συνέδριο της Ρουμανίας φτάνει σε επίπεδο και μεθοδολογία αντίστοιχο με αυτό του ευρωπαϊκού. Και λόγω των ε, καθηκόντων μου ενεπλάκην και στην αναδιάρθρωση του ελεγκτικού συνεδρίου και στην μια διαδικασία διαρκούς προσωπικής επιμόρφωσης. Έτσι, προχωρούμε στην ενίσχυση και εδραίωση των θεσμικών ικανότητων για έλεγχο και επαλήθευση των δημοσίων οικονομικών. Συνέλαβα λοιπόν την ιδέα της προαγωγής της πολιτικής, της οικονομικής, ε, του οικονομικού ελέγχου και τη διαχείριση των ανθρωπινών πόρων. Επί 17 έτη είχα την καθοδήγηση ελεγκτικών δράσεων σχετικών με τη ε, κονδύλια για τις περιφερειακές δομές του Λεκτικού Συνεδρίου για επαληθεύση των επενδύσεων και των δημοσίων προμηθειών. Ως Γενικός Γραμματέας ανέλαβα την προαγωγή της λειτουργίας κατά τρόπο αποτελεσματικό και παραγωγικό της ομάδας μου, της εχειριστικής. Μπόρεσα να αναβεθμίσω τις προσωπικές μου δεξιότητες, ώστε να έχω μια πανοραμική εικόνα της λειτουργίας ενός ελεκτικού συνεδρίου, που πρέπει να είναι ανεξάρτητος, αξιόπιστος και υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας οργανισμός, ο οποίος επαληθεύει τα δημοσιοοικονομικά. Ως άρδοτος ε, υπαλληλό στο ελεκτικό συνέδριο, του οποίου μάλιστα το προϊόν εργασίας από το 1994 έως το 2013 όλα αυτά τα συναπτά έτη ε, έχει τύχει επιβεβαίωσης και επικρότησης από όλες τις αντίστοιχες ε, πολιτικές αρχές, μπορώ νομίζω να παρουσιάσω μία ε, εικόνα, ένα βιογραφικό υψηλού επαγγελματισμού, αποδοτικότητας και ανεξαρτησίας. Τώρα και με την ελπίδα ότι θα υποστηρίξει η σύστασή σας την δική μου ψηφιότητα, θα ήθελα να καταστώ συνομιλητή σας, συνδιαλεγόμενος, εν ώψη μια στενή συνεργασία με τα μέλη τη Επιτροπή σα, που πιστεύω ότι θα μα επιτρέψει να συλλέξουμε τι απόψεις, προτάσει, ιδέε σα για τη λειτουργία του οργανισμού του Λακτικού Συνεδρίου. Με στη διάθεσή σα ανά πάσα στιγμή το θελήσετε και είμαι πεπισμένος ότι οι δραστηριότητε του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν μπορούν να ολοκληρωθούν επιτυχώς χωρίς την συνεργασία και την στενή διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο παρακολουθεί την υλοποίηση στο κομμάτι της διαδικασίας που του αντιστοιχεί της εκτέλεσης του προπολογισμού. Και επίσης σκοπεύω να ε, εφαρμόσω τις συστάσεις και προτάσεις που έχει διατυπώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ελεκτικό Συνέδριο προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να γίνει διόρθωση των διαπιστωθέντων σφαλμάτων. Και πριν ολοκληρώσω, θα ήθελα να σας βεβαιώσω ότι σημεριζόμαστε και εσείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου ένα έργο πολύ σημαντικό, την διασφάλιση δηλαδή της απρόσκοπτης, αποτελεσματικής, διαφανούς και άψογης διαχείρισης του ευρωπαϊκού ε, προϋπολογισμού, των χρημάτων δηλαδή από το, που καταβάλει ο Ευρωπαίος Προλογούμενος, ιδιαίτερα σε μια περίοδο δύσκολη, με πολλαπλές κρίσεις όπου χρειάζεται να ε, εδρεωθεί ακόμη περισσότερο κάθε είδους πλεονέκτημα που μπορεί να προσφέρει ο Ευρωπαϊκός Προπολογισμός για τον πολίτη ως μέρος και ως όλων. Σας ευχαριστώ πολύ και περιμένω με ενδιαφέρον τις ερωτήσεις και σχόλια που ενδεχομένω έχετε. Σας ευχαριστώ θερμά και τώρα παρακαλώ η κυρία Ζέντερ να λάβει το λόγο πρώτη, μια και το ζήτησε. Eh, ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, κύριε Πουφάνη, να σας καλωσορίσω στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε ενώπιον μας κάποιον ο οποίος ε, συμμετείχε ενεργά σε ελεγκτικό συνέδριο χώρας για 20 χρόνια ε, περίπου μάλιστα. Ε, είστε κάποιος λοιπόν στον οποίο δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε πώς λειτουργούν τα ελεκτικά συνέδρια και εγώ επειδή ακριβώς έχετε και μακρά πείρα θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση σχετικά με την αναδιοργάνωση που χρειάστηκε να κάνετε το 2003 ε, στο ελεγκτικό συνέδριο της Ρουμανίας προκειμένου να εξυγχρονιστεί και να προσαρμοστεί ε, στις παραδόσεις και στα κριτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσατε ίσως να μας εξηγήσετε λίγο καλύτερα με ποιο τρόπο αναλάβατε το συγκεκριμένο καθήκον και τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε και τι διδάγματα θεωρείτε ότι αντλήσατε, τα οποία θα μπορούσατε ίσως να σας βοηθήσουν ε, στο ελεγκτικό συνέδριο. Θα ήθελα επίσης ε, να σας ρωτήσω και το εξής. τις ε, συστάσεις ε, και στις πιθανές συμβουλές αναφέρεστε στην περίπτωση της ε, Ρουμανίας και της συνεργασίας και θεωρείτε ότι αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα για το μέλλον και για τις εθνικές ελεγκτικές αρχές. Διότι το σημαντικό πρόβλημα για μας δεν είναι μόνο ο έλεγχος του ευρωπαϊκού προπολογισμού αλλά κυρίως ο έλεγχος από πλευράς κρατών μελών, ε, τον οποίο θα πρέπει να κάνουν τα ίδια τα κράτη-μέλη με αποτελεσματικό τρόπο σε εθνικό επίπεδο και να μπορέσουν έτσι να κινητοποιηθούν και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Ε, Αναφερθήκατε στα προενταξιακά ταμεία στη Ρουμανία και θεωρείτε ότι αυτό είναι καλό παράδειγμα. Θεωρείτε ότι το παράδειγμα αυτό θα μπορούσαμε ίσως να το χρησιμοποιήσουμε και να το εφαρμόσουμε και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και επίσης από την πείρα σας Ποια στοιχεία μπορέσατε να χρησιμοποιήσετε, με ποιο τρόπο δηλαδή οι γνωμοδοτήσεις του Ρουμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου χρησιμεύσαν και χρησιμεύουν για να καταπολεμήσετε οποιονδήποτε κίνδυνο ή ένδειξη, απάτηση, διαφθοράς. Ε, διότι όπως γνωρίζετε εμείς στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού επανειλημμένως ε, έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της διαφθοράς ε, και την κατάσταση στη Ρουμανία εν γέννη. Και τέλος, ε, μία ερώτηση σχετικά με τη διαβίου μάθηση, διότι εσείς είστε ένα εγνωσμένο κύριος μέλος, αυτό ακριβώς που πρεσβεύουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν σταματάτε ποτέ να ε, βελτιώνετε την ε, εκπαίδευσή σας. Ε, υπάρχουν εδώ συμμετοχή σε διάφορα σεμινάρια, στο Βερολίνο και ούτω καθεξής λαμβάνετε πτυχίο στο Πανεπιστήμιο στο Γαλάτσι, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, διότι έχουμε μια συνάδελφο που έχει σπουδάσει εκεί και πολλές φορές έχω πάει στην πόλη σας, ε, στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Λογιστικών και θα ήθελα να ξέρω ε, τι σας έκανε το 2008 να θεωρήσετε ότι θα πρέπει να ε, σπουδάσετε και άλλα πράγματα και να λάβετε και το πτυχίο Οικονομικών Επιστημιών και να προχωρήσετε την εκπαίδευσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να απαντήσετε αν θέλετε αμέσως. Σας ευχαριστώ πολύ. Στην πρώτη σας ερώτηση θα έλεγα ότι όσον αφορά την επανοργάνωση του ελεκτικού συνεδρίου στην Ρουμανία και σε σχέση με διάφορες πρακτικές που ισχύουν εκεί. Όσον αφορά τη δραστηριότητα μετά το 2003, από το 2003 δηλαδή και πέρα, οι παρόντες μέλη του Ελεκτικού Συνεδρίου εκείνη την εποχή αντικαταστάθηκαν και το 2005 η συνταγματική μεταρρύθμιση οδήγησε και σε κάποιες άλλες αλλαγές. Πρέπει να σας πω ότι διάφορα μέλη του τότε ελεγκτικού συνεδρίου αντικαταστάθηκαν και μετά την αποχώρησή τους. Ιδιαίτερα αναφέρομαι εδώ στους δικαστές. Το ελεγκτικό συνέδριο βρέθηκε σε μία φάση αρκετά δύσκολη αναδιάρθρωσης και κάποιες υποθέσεις οι οποίες ε, είχαν φτάσει ε, στη δικαιοσύνη. οδήγησαν στην εκπροσώπηση του συνεδρίου κάτι που δεν ήταν πάντα προς ε, του θεσμού. Ο έλεγχος ουσιαστικά έγινε από μέλη του συνεδρίου με την πλαισίωση βεβαίως κάποιων νομικών συμβούλων. Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι κάποιες από τις υποθέσεις δεν προχώρησαν ή άλλες τελικά δικάστηκαν σε άλλα δικαιοδοτικά όργανα, σε άλλα δικαστήρια. Παρ' όλα αυτά πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν χώρες όπως η Ισπανία και η Γαλλία, υπάρχουν αντίστοιχα όργανα τα οποία μπορούν να αναλάβουν αυτές τις υποθέσεις. Και η κατάσταση είναι πολύ πιο απλή. Όταν είχα πάει στη Μαδρίτη μπόρεσα να επισκεφτώ αυτό το το δικό τους όργανο. Πρέπει να σας πω ότι έχω στενές επαφές με συναδέλφους από την Μαδρίτη, από το Ηνωμένο Βασίλειο και μάλιστα αποφάσισα να επανέλθω στο Πανεπιστήμιο της πόλης μου, γιατί θεωρώ ότι αυτή η επαγγελματική κατάρτιση είναι πάρα πολύ σημαντική για την σταδιοδρομία μου. Με αυτόν τον τρόπο μπορώ να καταλάβω πολύ καλύτερα περί τίνος πρόκειται και πώς μπορεί κανείς να δεκτερεώσει έναν τέτοιο έλεγχο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πούφαν. Θα δώσω το λόγο τώρα στους συναδέλφους που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις. Ο κύριος Ιβάν. Νομίζω πρέπει να πάμε ανάλογα με την δύναμη των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Οντί είναι πριν από εσάς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να σας καλωσορίσω κύριε Πούφαν και να σας κάνω και τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση αφορά τις αρμοδιότητες, τις δεξιότητές σας. Η συνθήκη προβλέπει ότι τα μέλη των εθνικών συνεδρίων είναι μπορεί να είναι υποψήφοι για τη θέση την οποία θέλετε να αναλάβετε ή, ή να έχετε κάποιες ε, ειδικέ ε, ε, κάποιες δεξιότητες, κάποια εμπειρία στον τομέα του ελέγχου. Καταλαβαίνετε ότι θα μπορέσετε από τη στιγμή που θα εκλεγείτε να συμμετάσχετε σε ένα συλλογικό όργανο ελέγχου να εφαρμόσετε και να υλοποιήσετε κάποιες διαδικασίες, κάποια διεθνή λογιστικά πρότυπα. να Αναρωτιέμαι λοιπόν αν τα γνωρίζετε, αν όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στην κατάρτιση που όπως μας είπατε είχαν πρόσφατα ή αν θα χρειαστεί κάποια συμπληρωματική κατάρτιση. Μπορείτε να μας πείτε αυτό το δίπλωμα που περάσατε πρόσφατα για να συμπληρώσετε τις γνώσεις σας στον ε, λογιστικό έλεγχο, τι ακριβώς περιεχόμενο είχε. Διαβάζω το βιογραφικό σας. Λέτε ότι υπάρχουν 42 ελεκτικά συνέδρια περιφερειακά στη Ρουμανία και ότι εσείς ήσασταν ο συντονιστής. Παίξατε έναν συντονιστικό ρόλο στον λογιστικό έλεγχο αυτό καθεαυτό ή σε διοικητική θέση ήσασταν. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς πώς λειτουργεί το ελεγκτικό συνέδριο της Ρουμανίας. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές ερωτήσεις έκανε κύριε Σοντή. Κύριε Πούφαν, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε κύριε Οντή για την ερώτησή σας. Θα ξεκινήσω με το πτυχίο μου. πτυχίο οικονομικών με ε, εξειδίκευση στη λογιστική στα πλαίσια της ε, συνεχούς ε, μάθησης, της διαβίου μάθησης πήγα σε προχωρημένη ηλικία να πάρω ένα δεύτερο πτυχίο. μας, μου θέσετε και την ερώτηση για τα ε, ελεγκτικά συνέδρια της Ρουμανίας και ε, εκεί να σας πω ότι εργάστηκα σε αρκετές ε, περιπτώσεις, σε διάφορους τομείς και σε κάθε περιφέρεια υπάρχει το ε, αντίστοιχο ελεγκτικό συνέδριο και φυσικά εκεί γίνεται έλεγχος ε, για τις κρατικές προμήθειες. Και φυσικά ως ελεγκτής ε, και διατάκτης είμαστε υπεύθυνοι για την επαλήθευση των ε, δημοσίων λογαριασμών και των εσόδων, λαμβάνοντας για παράδειγμα έστω ότι δημιουργούνται υποδομές, ε, ένα αθλητικό κέντρο ή ένα σχολείο. Εγώ ήμουν υπεύθυνο της ομάδας που διενεργούσε τον έλεγχο και από το 1994 στο 2004 ε, συμμετείχα σε αυτή τη διαδικασία ε, επαλήθευσης των ε, δημοσίων λογαριασμών, έκανα τον έλεγχο των έργων, τα λογιστικά στοιχεία, τα οικονομικά στοιχεία, τον οικονομικό φάκελο, τι γίνεται με τα έργα τα οποία κατασκευάζονται, τι προτείνεται, ποιες προτάσεις υποβάλλονται και φυσικά γινόταν και ένας έλεγχος προκειμένου να επαληθεύσουμε ότι έγινε σωστά η δαπάνη. Πρόκειται για μία απαλλαγή ουσιαστικά ε, σε επίπεδο κάθε περιφερειακού ελεκτικού συνεδρίου των 42 ελεγκτικών συνεδρίων της Ρουμανίας. Και από εκεί και πέρα υπήρχε ένα σύνολο εκθέσεων, ε, υπήρχαν 42 περιφέρειες φυσικά και επικεντρωνόμασταν ε, σε κάποιες περιπτώσεις στις πιο σημαντικές δαπάνες και ε, κοιτούσαμε από πλευράς ελεγκτικού συνεδρίου αν έγιναν σωστά τα πάντα. Επρόκειται για έναν έλεγχο και όταν υπήρχε πρόβλημα για τα έγγραφα, την παρουσίαση, τη δομή, την ε, ελεγκτική ομάδα ή οποτεδήποτε υπήρχε κάποια αμφιβολία, ο Υπουργός μπορούσε κάλλιστα να ε, μεταβεί επιτόπου προκειμένου να διαπιστώσει ε, τι συμβαίνει. Και ως ε, κύριος διατάκτης, εγώ ήμουν υπεύθυνος για τη διεξαγωγή του ελέγχου και μπορούσα να κάνω και επιπλέον ε, ε, επαληθεύσεις και ελέγχους. Και φυσικά έπρεπε στη συνέχεια να υποβληθεί μια τελική έκθεση και όπως κάνει και ο Γενικός Γραμματέας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να παρουσιάζεται η έκθεση αυτή στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στη συνέχεια ε, περνούσαμε στο θέματα της εκτέλεσης του προπολογισμού και φυσικά ε, από την αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου της Ρουμανίας. Μου θέσατε και μία ερώτηση και με ρωτήσετε τι θα έκανα εάν διοριστώ. στο αρμόδιο τμήμα του ελεγκτικού συνεδρίου στο Λουξεμβούργο Ο συνάδελφος τον οποίο θα αντικαταστήσω ασχολείται με θέματα μεταφορών και ενέργειας είναι στο αρμόδιο τμήμα και εάν ε, μου ανατεθούν αντίστοιχα καθήκοντα από τον πρόεδρο του ελεκτικού συνεδρίου, είναι ένας τομέας στον οποίο έχω ε, μακρά πείρα και θεωρώ ότι θα μπορώ να διεξάγω τα καθήκοντα τα οποία... Ε, ευχαριστώ πολύ. Μου ζητάτε. Ο κύριος Σιβάνα το λόγο. σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ιδιαίτερα για τη φροντίδα που ε, χαρακτηρίζει την προετοιμασία σας. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο προτέρημα για κάθε στάδιο της ζωής και ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε υποβληθεί σε επιθέσεις πρόσφατα, ξέρω ότι δεν ήταν τεκμηριωμένες και στο συγγνώμη εκ μέρου των συναδέλφων συμβαίνουν και πράγματα στη Ρουμανία και δεν έβαλαν προσωπικό εναντίον σας αυτές οι κατηγορίες, αλλά Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να πείσουμε την κυρία Μακοβέη, την συνάδελφο, να σας υπερψηφίσει και εκείνη. Έχω όμως μια πιο συγκεκριμένη ερώτηση. Οι εμπειρίες σας, οι δραστηριότητες σας είναι καθαρά διοικητικού χαρακτήρα. Δώσατε απαντήσεις στα υπόλοιπα ερωτήματα, αλλά εγώ έχω να επιμείνω σε κάτι σχετικό με το δημοσιονομικό έλεγχο, διότι έχουμε δει υποψηφιότητε στην Επιτροπή μα και συναδέλφων και άλλων που δεν είχαν μεγάλη εμπειρία ως προς το δημοσιονομικό έλεγχο, αλλά που εν τέλει ενεκρίθη η υποψηφιότητά τους από τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κατέστησαν έτσι μέλη του Ελεκτικού συνεδρίου. Ήθελα λοιπόν να μου πείτε αν έχετε κάποια συγκεκριμένη εμπειρία από δημοσιονομικό έλεγχο, κάτι συγκεκριμένο από τη δραστηριότητά σας και επίσης θα ήθελα να μας πείτε τα θεσμικά όργανα στα οποία έχετε εργαστεί, τι ζητήματα σχετικά με την απαλλαγή έχετε αντιμετωπίσει. Υπήρχε ένα, μια αντίσταση από, το, από την ε, δεξιά του PDL, του κόμματος PDL, ε, στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο τι έγινε τελικά, δώσανε την έγκρισή τους για την απαλλαγή ή όχι σε εκείνη την περίπτωση. Ο κύριος Πουφάνη. σας ευχαριστώ πολύ. Για το δημοσιονομικό έλεγχο, όπως έλεγα και νωρίτερα. Έχω πειρα 19 ετών στο ελεγκτικό συνέδριο της Ρουμανίας. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πολλές ήταν οι φορές όπου έλαβα μέρος σε δραστηριότητες ελεγκτικές Έχω διεξαγάγει δημοσιονομικού ελέγχους, το επαναλαμβάνω με επιφάσεως. Οι δύο θέσεις που είχα το 1994 ω ανώτατο αξιωματούχο και από το 2002 τον Ιούλιο ω Γενικό Γραμματέας ήταν θέσεις που κατέλαβα κατόπιν διαγωνισμού και ξέρετε όταν διορίζεται σε Υπουργείο Γενικός Γραμματέας διορίζεται με διαφορετικού όρου, τον διορίζει ο Πρωθυπουργό. Εγώ όμω πέρασα διαγωνισμό. Και θα ήθελα επίση να επισημάνω ότι και οι σπουδέ μου στο Πανεπιστήμιο του Γαλατσί είναι σχετικέ, είναι οικονομικέ. Έχω ε, ειδικότητα τα λογιστικά. Πρόκειται για ένα ανεγνωρισμένο πανεπιστήμιο. Μπορώ να σας διαβιβάσω αν θέλετε και το πρωτότυπο των διπλωμάτων μου για επαλήθευση. Έχω επίσης ε, διδαχθεί την ε, διαδικασία επαλήθευσης λογαριασμών στο Πανεπιστήμιο, στις σπουδές μου. Έχω σπουδάσει τόσο στη Ρουμανία όσο και στο εξωτερικό. Και πιστεύω ότι είμαι σε θέση να εργαστώ στο ελεγκτικό συνέδριο το ευρωπαϊκό, ότι έχω τα κατάλληλα προσόντα. Τώρα, όσον αφορά την απαλλαγή, τη διαδικασία απαλλαγής για την εκτέλεση του προπολογισμού, στις δραστηριότητε μου ως, γενικού γραμματέως είχα αυτή την διαδικασία, την ε, έζησα αρκετές φορές, εμφανίστηκε δηλαδή ο γενικός γραμματέας ενώπιον του ε, Κοινοβουλίου, παρουσιάζει τον, την έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου σε σχέση με τις ε, δαπάνες από τον Εθνικό Προπολογισμό. Εάν υπάρξουν ερωτήσεις προς το ελεγκτικό συνεδρίο από την Ολομέλη, αν υπάρξουν παρατηρήσεις, υπάρχει, προβλέπεται η δυνατότητα της διόρθωσης στην έκθεση, αλλά τέτοιου είδους ζήτημα δεν εμφανίστηκε ποτέ στη δική μου στοιδρομία. Έτσι λοιπόν, στη συνέχεια αποστέλλεται το κείμενο στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού της Γερουσίας της Ρουμανίας, η οποία έχει την ε, απαλλαγή και επαλήθευση, έγκριση της εκτέλεσης των προϋπολογισμών. Αυτή είναι η διαδικασία. Τα 11 χρόνια όπου είχα τη, κατήχα τη θέση του Γενικού Γραμματέα δεν αντιμετώπισα ποτέ αντίδραση ως προς ε, τις εκθέσεις για δημόσιες προήθειες ή δραστηριότητες γενικά του Γενικού Γραμματέα ε, που κατήχα αυτά χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μίλντερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εξή. Ένα από τα καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι κάθε χρόνο να καταθέσει τη έκθεση για την κατάσταση ε, των πεπραγμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που ονομάζουμε DAS, δηλαδή δήλωση αξιοπιστία, που έχει ε, παρουσιαστεί αρκετές χρονιές αρνητικό, τώρα έχουμε μια κάποια βελτίωση, αλλά αν κοιτάξει κανείς, ε, και αν, κάνει κανείς μια αναδρομή, βλέπει μια βελτίωση σταδιακή, ελαφρά έστω. Θα θέλατε λοιπόν να μας κάνετε κάποια πρόταση για το πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση ως προς τη θετική δήλωση αξιοπιστίας και να μας δώσετε κάποιες ε, ενδεχομένως δικές σας εμπειρίες από τη Ρουμανία, αν υπάρχει αντίστοιχο σύστημα. Και τι είδου τάσεις είδατε τα τελευταία χρόνια με το δημόσιο προπολογισμό, με το προπολογισμό στη Ρουμανία. Απάντηση. Σας ευχαριστώ κύριε Πουφάν. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μιούλτερ για την ερώτηση. Όπως γνωρίζουμε, η δήλωση εξοπιστίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν τα τελευταία 17 χρόνια δυστυχώς αρνητική. Σημαίνονται δηλαδή κάποιες αντιφάσεις μεταξύ της χορήγηση της δήλωση προς την εκτίση εξέταση των ε, λογαριασμών και του γεγονότος ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολυετής, αυτή η απόκληση σημαίνει προβλήματα. Υπάρχει επίσης προ το σφάλματος που καταγράφεται στη δήλωση. Το οποίο είναι πιο σημαντικό, πιο υψηλό. από θα έπρεπε να έχουμε στην ε, πραγματικότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν μπορεί να έχει επιβάλει πολύ σκληρέ κυρώσει σε ορισμένε περιπτώσει. Πλην όμω διαπιστώνουμε ότι ορισμένε χώρε δεν είναι σε θέση να ε, αρθούν στο ύψο των απαιτήσεων τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίση βλέπω ότι ρωτάτε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στη Ρουμανία. Εάν υπάρχει αντίστοιχη ε, δήλωση εξοπιστίας για το Ρουμανικό Ελεκτικό Συνέδριο. Να σας πω, για τον γενικό προϋπολογισμό, τον ενοποιημένο προϋπολογισμό, τέτοιου είδους δήλωση εξοπιστίας δεν προβλέπεται. Αλλά σε κάθε χωριστό τμήμα, φερειπίν κοινωνικές ασφαλίσεις, προϋπολογισμός της γενικής κυβέρνησης και το καθεξής, έχουμε αντίστοιχα δήλωση εξοπιστίας στη Ρουμανία. Ο πρόεδρος ευχαριστώ. Κυρία Κρέσλε, σας ευχαριστώ. Χαίρομαι που μπορούμε να τα ξαναπούμε κύριε Πουφάν. Θα ήθελα για όσους παρακολουθούν από τα κράτη-μέλη να επισημάνω ότι είναι πολύ καλό να έχουμε υποψηφίους κάποτε που να μην χρειάζονται. Συνοδεία. Κύριε Ποφάν, πολλοί σας γνωρίζουν εσάς και στην Ρουμανία και αλλού πολύ καλά. Για το σημείο 10, στην ερώτηση καλύτερα 10, όπου βλέπουμε τι είδου ε, προστιθέμενη αξία μπορεί να προσφέρουν ε, οι δημοσιονομικοί έλεγχοι. Πρόκειται για ένα σημαντικό ζήτημα, ε, δημοσιονομική έλεγχη επιδόσεων έλεγχος επιδόσεων, performance audits, και με ποιους τρόπους θα έπρεπε τα πρόσματά του να σηματώνονται στις ε, διαδικασίες του management. Εδώ λοιπόν βλέπω ότι η απάντησή σας είναι μια αντιγραφή της σελίδας 26 ε, του, ε, της εκθέσεως του 1998. Copy-paste ακριβώς. Ερωτώ λοιπόν, έχετε δική σας γνώμη ή απλώς αντιγράφετε κάποιο κείμενο και πώς θα εξηγήσω ότι μας κάνετε ένα copy-paste της εκθέσεως του Ρουμανικού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και πώς είναι δυνατόν πάλι να διαπιστώνουμε ότι δεν έχει και τόσο πολύ καλά υλοποιηθεί όλο αυτό το σύνολο των αποτελεσμάτων. Κύριε Πουφάνη, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Γκρέσλε, για την ερώτησή σας. Όσον αφορά την απάντησή μου στην ερώτηση 10, πρέπει να σας πω ότι όσοι εργάζονται στο ελεγκτικό συνέδριο της Ρουμανίας έχουν συμμετάσχει πλιστάκης σε προετοιμασία των προδιαγραφών για προγράμματα δημοσιονομικών ελέγχων ή άλλων είδων ε, audit, έλεγχο επιδόσεων κτλ. Χρησιμοποίησα λοιπόν ένα κείμενο γιατί η δράση μου πραγματικά είναι μια δράση που συμβαδίζει με όλη αυτή την διαδικασία. Ένας ε, άνθρωπος ο οποίος εμπλέκεται σε τέτοιους ε, ελέγχους θα πρέπει να μπορεί να διαπιστώσει, θα πρέπει να έχει και την δυνατότητα να διαισθανθεί ορισμένα πράγματα και νομίζω ότι ο ρόλος μου και η δράση μου σε πολλούς δημοσιονομικούς ελέγχους, ελέγχους επιδόσεων, μου έχουν δώσει μια τέτοια εμπειρία και θεωρώ και όλος ότι έχω και κάποιες ηγετικές ικανότητες όσον αφορά αυτούς τους ελέγχους. σε ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μακοβάη. Thank you, President. Um... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν ε, κατάλαβα από την απάντησή σας γιατί πρόκειται περί του ακριβώς ίδιου κειμένου με αυτό που υπάρχει στην έκθεση. Ακριβώς το ίδιο κείμενο. Αντιγραφή. Τώρα, όσον αφορά την χρήση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ε, καταλαβαίνετε ότι εδώ είναι καθοριστικό το πώς το ελεγκτικό συνέδριο θα προασπιστεί τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, πώς ε, μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι η χρήση τους είναι ορθή. Αλλιώς καταλαβαίνετε αποδυναμώνουμε το ελεγκτικό συνέδριο και μειώνουμε και την αξιοπιστία του. Θα ήθελα λοιπόν, και εδώ απευθύνομαι σε όλους τους συναδέλφους, να ζητήσω από όλους να κοιτάξουν τα απτά γεγονότα και όχι την ιδεολογία. Γιατί ο λόγος για τον οποίο επιλέγουμε κάποιον για να βρεθεί στο ελεγκτικό συνέδριο πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία και όχι σε ιδεολογικές προσεγγίσεις. Λέτε ότι το 2011 πήρατε πτυχίο από το Πανεπιστήμιο του Καλάτσι, ότι ήσασταν δηλαδή από το 2008 στο 2011 σπουδάσατε, ήσασταν φοιτητή στο Πανεπιστήμιο αυτό. Την ίδια ώρα ήσασταν Γενικός Γραμματέας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Βουκουρέστι. Καταλαβαίνετε ότι η απόσταση μεταξύ του Πανεπιστημίου και του Βουκουρέστι και της πόλης του Βουκουρέστη υπάρχουν 250 χιλιόμετρα απόσταση. Είναι πολύ δύσκολο να κατανοήσω λοιπόν πώς μπορείτε εσείς να είστε ταυτόχρονα και στο Πανεπιστήμιο και στο Βουκουρέστη στο ελεγκτικό συνέδριο. Πρόκειται, επαναλαμβάνω, για δύο πόλεις οι οποίες απέχουν 250 χιλιόμετρα. Και πώς καθημερινά κάνατε αυτές τις διαδρομές. Εγώ κοίταξα το, την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου σας και είδα ότι τα μαθήματα είναι από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή. Πώς μπορούσατε λοιπόν να ήσασταν ταυτόχρονα σε δύο σημεία. Δεύτερη ερώτηση. Που αναφέρεται στα ίδια χρόνια. Ουσιαστικά είστε πτυχιούχος όχι δημοσιονομικού ελέγχου, αλλά του λογιστικού τμήματος του Πανεπιστημίου αυτού. Θεωρείτε ότι έχετε τις απαραίτητες δεξιότητες και προσόντα στον τομέα του ελέγχου. Από ό,τι βλέπω, πήρατε τη βάση. Ο βαθμός σας είναι 5 στα 10. Εξάλλου και σε πολλά άλλα μαθήματα ο βαθμός σας είναι η βάση. Βλέπω στη σελίδα 4 του βιογραφικού σας ότι ήσασταν από τους 183 σπουδαστές ο 161ος, δηλαδή μεταξύ των τελευταίων φοιτητών. Αυτή λοιπόν η έλλειψη επιδόσεων, η οποία είναι τεκμηριωμένη, δείχνει ότι ίσως ε, δεν είστε κατάλληλος. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος Πούφαν. Σας ευχαριστώ κυρία Μακοπαή για τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, όσον αφορά το Πανεπιστήμιο του Δούναβη, το Καλάτη, όντως παρακολούθησα μαθήματα από το 2008 στο 2011 και πρέπει να σας πω ότι την ίδια αυτή η περίοδο ίσως σήμερα έχει αλλάξει η κατάσταση αλλά τα μαθήματα τότε ήταν Παρασκευή και Σάββατο τότε, επειδή δεν υπήρχαν πολλοί σπουδαστέ, υπήρχε μεγάλη ευελιξία στη διοργάνωση των μαθημάτων και δεν ήταν υποχρεωτική η παρουσία στα μαθήματα. Γι' αυτό και ε, μπορώ να σας ε, εξηγήσω αυτό το πτυχίο. Στα 53 μου χρόνια πήρα το πτυχίο γιατί ήθελα να συμπληρώσω τις σπουδές μου, να προσθέσω αυτή την κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση και όσον αφορά τους βαθμούς μου αντιστοιχούν στην προσπάθειά μου. Έκανα ό,τι μπορούσα. Μπορεί κάποιος ε, να σχολιάσει βεβαίως τους βαθμούς μου σε κάποια μαθήματα. Αλλά τι να σας πω, ήμουν 50 53 ετών και πρέπει να σας πω ότι οι επιδόσεις μου δεν ήταν στο ύψος ε, ενός σπουδαστή 20 ετών. Θα κάνω ό,τι μπορώ, θα συνεχίσω να τελειοποιούμε και να συμπληρώνω την κατάρτισή μου έτσι ώστε να φτάσω στο ύψος ε, το οποίο σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι έχουμε ολοκληρώσει την ακρόαση αυτή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, έχετε κάποιες ερωτήσεις συμπληρωματικές, δεν βλέπω κανέναν. Θα δώσω το λόγο πάλι στην εισηγήτρια, αν το επιθυμεί. Sí, gracias, presidente. Sí. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη κύριε αν συνήθως εδώ στην Επιτροπή μας δεν ασχολούμαστε με ανώνυμες καταγγελίες που έχει αποστείλει κάποιος μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μάλιστα έχει φτάσει και στα μηνύματα της κυρίας Μακοβέη. Ζητώ συγγνώμη, δεν είναι η συνήθις διαδικασία που ακολουθούμε. Ασχολούμαστε με έγγραφα τα οποία είναι υπόγραφα και ε, αποδεικνύονται και κάπου. Ήθελα απλώς να υπενθυμίσω στην κυρία Μακοβέη ότι ούτε και ο Αλμπέρτ Αϊνστάιν ήταν και ο καλύτερος μαθητής στην τάξη. Και εγώ ενώ εργαζόμουν έκανα και μαθήματα νομικής ε, και χρησιμοποιούσα τη δυνατότητα που έχουν ε, οι καθηγητές πανεπιστημίου να δείχνουν μια κατανόηση. Κάποιοι οι οποίοι είναι εργαζόμενοι και ταυτόχρονα φοιτητές ε, έχουν μια κάποια βοήθεια, τους διευκολύνουν και οι καθηγητές και οι συμφοιτητές τους. Δεν καταλαβαίνω που έγινε το πρόβλημα και γιατί αυτό θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα και δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι είναι και ε, το Πανεπιστήμιο Ντανούμπιο στο Γαλάτσι είναι πανεπιστήμιο ε, δεύτερης κατηγορίας ε, γιατί διευκολύνει τους φοιτητές του. Θα ήθελα να υπενθυμίσω και πάλι ότι συνήθως δεν έχουμε υποψηφίους που να έχουν τόσο μεγάλη πείρα σε εθνικό ελεγκτικό συνέδριο, το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι ακριβώς προσπαθούμε να ε, δημιουργήσουμε μια νέα σχέση με τα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε στον έλεγχο των προπολογισμών τους και είναι ένας από τους λίγους υποψηφίους που είχαμε εδώ που γνωρίζει και τις διαδικασίες ε, διαχείρισης ε, ε, και μάλιστα τις έχει χρησιμοποιήσει επανειλημμένως και για τόσα πολλά χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι σε αυτή την περίπτωση καλύπτονται οι βασικές μας απαιτήσεις και θα ήθελα να μην υπενθυμίσουμε εδώ και το βιογραφικό σημείωμα άλλων υποψηφίων που έχουμε εγκρίνει στο παρελθόν, που δεν είχαν τόση πείρα και δεν μας δημιούργησαν κανένα πρόβλημα. Καταλαβαίνω ε, βέβαια ε, ότι ορισμένοι μπορεί να θεωρούν πρόβλημα, αλλά ε, ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχίζει να σπουδάζει ενώ εργάζεται δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα. Το 2008 άλλωστε δεν ήταν καν υποψήφιο για το ελεκτικό συνέδριο και δεν καταλαβαίνω γιατί δημιουργείται τέτοιο θέμα με το πτυχίο σας από το Πανεπιστήμιο στο Γαλάτσι, το οποίο ούτως ή άλλως έγινε και αποδεκτό από το αρμόδιο Υπουργείο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε και σε αυτή την ερώτηση. Α, με συγχωρείτε όμως. Και η κυρία Μακοβέη θέλει το λόγο πάλι. Ας ξεκινήσουμε με αυτήν πρώτα. Παρακαλώ. Πρόεδρε, μια και η κυρία Γιάλα Σέντερ ε, ανέφερε το όνομά μου. Διατυπώνω τις ερωτήσεις που θεωρώ ενδιαφέρουσες. Για όλους μας, για όλες τις πολιτικές ομάδες διότι θέλουμε να ενισχύσουμε τον, το, το θεσμό του ελεγκτικού συνεδρίου. Δεν έχει σχέση αυτό με την εσωτερική πολιτική. Τις προτάσεις κάνει η κυβέρνηση. Δεν έχει θέμα αυτό, δεν έχει σχέση με μικροπολιτικές. Μόνο με ικανότητες. Αλλά ρωτώ, συγκρίνατε τώρα τον κύριο που με τον κύριο Αϊνστάιν. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για την ε, παρέμβαση κυρία πρόεδρε. Δεν έκανα καμία σύγκριση, απλώς ήθελα να πω ότι αυτό που είπατε εσείς ε, για το, την παρουσία στα μαθήματα ως απλή και μόνο απόδειξη για καλή παιδεία δεν είναι ε, απαραίτητο. Σας έδωσα απλώς το πιο γνωστό παράδειγμα για να γνωρίζουν όλοι ότι υπήρχαν μαθητές οι οποίοι ναι μεν δεν συμμετείχαν στα μαθήματα ε, και μπορούν κάλλιστα να λάβουν το πτυχίο τους και να προχωρήσουν τη σταδιοδρομία τους. Και απλώς είπα ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και ότι ο κύριος που φαν ήταν εργαζόμενο εκείνο το διάστημα. Ja, vielen ευχαριστώ. Και τώρα, για να ξεκινήσω εγώ, ο Άλμπερτ Άινσταϊν, ε, από ό,τι γνωρίζουμε, έλαβε βραβείο Νόμπελ για την θεωρία τη σχετικότητα. Ε, να δούμε τώρα εάν θα μπορέσει να αναπτύξει μια νέα θεωρία σχετικότητα στο ελεγκτικό συνέδριο Εάν θα μπορέσει δηλαδή να κάνει την ε, ρήξη αυτή στα δημοσιονομικά, στο δημοσιονομικό έλεγχο, ώστε να μπούμε σε μια νέα εποχή. Κύριε Πουφάν, μπορείτε να δώσετε απαντήσεις σε όποια ερώτηση ενδεχομένω έχει μείνει εκκρεμή, εάν το επιθυμείτε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Θα ήθελα να πω ότι Έχω όλα τα πρωτότυπα των πτυχίων μου. Όποιος θέλει είναι στη διάθεσή του. Πολύ ευχαριστώ να τα καταθέσω στην Επιτροπή σας. Πιστεύω ότι τα καθήκοντά μου πάντοτε τα έχω επιτελέσει με υψηλό πνεύμα επαγγελματικότητας και κύρους. Και όποτε έλαβα μέρος σε διεθνείς συνεδριάσεις στη Ρουμανία της στο εξωτερικό, είτε σε διμερείς είτε σε πολυμερείς συνεδριάσεις και επαφές με ε, προέδρους ελεκτικών συνεδρίων της Ευρώπης, της Ασίας, των ΗΠΑ πάντοτε, πάντοτε, και μπορώ να σας το πω αυτό, προσπαθούσα και προσπαθώ να δείχνω αποτελεσματικότητα και να παρακολουθώ με ιδιαίτερη προσοχή τον τρόπο εκτέλεσης του προπολογισμού, το πώς δαπανώνται τα δημόσια, το δημόσιο χρήμα. Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες και συντονιστικές συνεδριάσεις και άλλες στην Ρουμανία. Έχω λάβει μέρος σε συνεδριάσεις όπου είχαμε ε, και στοιχεία για τους υποψηφίους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα είμαστε στο τέρμα αυτής της δημόσιας ακρόασης. Ευχαριστώ κύριε Πουφάν για την παρουσία σας, για τις, απαφίες, για τις απαντήσεις σας ερωτήσεις και τώρα θα συνεχίσουμε και κλεισμένο των θυρών. Ευχαριστώ. Okay. Let's see. I don't. I, I don't doubt. Okay. So, um, ladies and gentlemen, I would kindly ask... Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ να μας ε, βοηθήσετε να βάλουμε μπρος το κομμάτι της συνεδριάσεως που γίνεται και κλεισμένο των θυρών όσο πιο γρήγορα. Yeah, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich Αγαπητοί συνάδελφοι, σα προτείνω να συνεχίσουμε με τη δημόσια συνεδρίαση. Λοιπόν, μόλις άκουσα ότι η κυρία Ντελάγκε δεν είναι εδώ, αλλά η κυρία Γκρέσλε είναι και θα την αντικαταστήσει η Σάξια. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε το λόγο στην κυρία Γκρέσλε, η οποία θα μιλήσει εξ ονόματος της εισηγήτριας. Θεωρώ πραγματικά ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Το θέμα της πολυγλωσσίας μας έχει απασχολήσει εδώ και πολύ καιρό και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις εξ ονόματος της εισηγήτριας όσον αφορά καταρχήν το, την πολυγλωσία έτσι ώστε ο καθένας, το κάθε μέλος του Κοινοβουλίου να μπορεί να εκφραστεί στην γλώσσα του. Η έκθεση αναφέρεται σε αυτά που έχουμε ήδη κάνει τα δύο τελευταία χρόνια. Ο Γενικός Γραμματέας έχει πάρει κάποιες αποφάσεις και βεβαίως έχουμε καταφέρει να περάσουμε κάποιες από τις αποφάσεις. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό βλέπουμε ότι προβλέπονται 10 εκατομμύρια λιγότερα για τις γλώσσες. Πρόκειται λοιπόν για μια πρόταση εξοικονόμησης, περικοπής των δαπανών, γιατί περί αυτού πρόκειται το θέμα της διερμηνίας και πώς θα κατενεμηθούν στη διάρκεια των συνεδριάσεων, ε, στις εβδομάδες, εβδομάδες του Στρασβούργου και τις αντιπροσωπείες. 10 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια έχουν ε, εξοικονομηθεί και αυτό θα φανεί εξάλλου στην απαλλαγή το 2013. Θα δείτε ακριβώς τους αριθμούς. Παραμένουν κάποια θέματα ακόμα εκρεμή, όπως η ακύρωση, η καθυστερημένη ακύρωση κάποιων συνεδριάσεων, πολύ σημαντικό κόστος αυτό και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς αυξάνεται ο αριθμός των συνεδριάσεων που ακυρώνονται τελευταία στιγμή. Χρειαζόμαστε περισσότερη λοιπόν ακρίβεια, χρειαζόμαστε εδώ κυρίως να ξέρουμε κάθε φορά πώς χρησιμοποιούνται αυτές οι δυνατότητες διερμηνίας, αυτά τα κονδύλια που προβλέπονται για τις γλώσσες και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα πρέπει πολιτικές ομάδες να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις. Θα έχουμε ένα νέο εργαλείο που θα είναι η διερμηνία μόνο εάν ζητηθεί να υπάρχει Interpretation on Demand. Θα υπάρξει και μια ειδική έκθεση για το θέμα αυτό, για την ε, διερμηνία, όπου θα ενημερώσουμε το θέμα αυτό και βεβαίως εδώ θα πρέπει το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή να έχουν κοινή θέση. Υπάρχουν κάποιες νέες προτάσεις, γίνεται μία ανάλυση εις βάθος για το τι είναι διερμηνία και κάποιες ε, προτάσεις, γιατί βεβαίως ε, οι γλώσσες και οι διερμηνίες συνεχίζουν να είναι μια σημαντική προσθέμενη αξία για την εργασία μας. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο. Συνάδελφοι, μέλη της Επιτροπής, δεν βλέπω κανένα να ζητάει το λόγο. Οπότε σας λέω απλώ ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 30 Μαΐου στις 12. Και θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω αυτό που είπε η κυρία Γκρέσλε εκ μέρους της εισηγήτριας. Το Κοινοβούλιο και μόνο το Κοινοβούλιο θα αποφασίσει πώς θα εργάζεται, με ποιο τρόπο θα υπάρξουν κάποιες εξοικονομήσεις, πώς θα χρησιμοποιηθούν κάποια κονδύλια. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ και θα πρέπει να το γνωρίζουν οι βουλευτές. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την υπηρεσία μετάφρασης και διερμηνίας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε εδώ να εργαστούμε. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. The reason for which we today. Mhm. Okay. Ja, wir sollten äh, aber die informieren, dass wir Η Φραντσέσκα μου ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, έχουμε προχωρήσει. Η γραμματεία με ενημερώνει ότι τον Απρίλιο, διάσκεψη των Προέδρων, πήρε κάποιες αποφάσεις για τις εκθέσεις για το επόμενο εξάμεινο. Και θα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις, θα πρέπει 1η Ιουνίου, αν δεν θέλουμε να χάσουμε κάποιες εκθέσεις, να αποφασίσουμε και να ορίσουμε τους εισηγητές. Συζητήσαμε με τους συντονιστές το θέμα κάποιων εκθέσεων Δεν ξέρω αν μπορούμε βεβαίως να ζητήσουμε δύο μήνες παραπάνω στην τελευταία συνάντηση των Προέδρων. Δεν νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Τώρα, εάν δεν χρησιμοποιήσουμε την ψηφοφορία του Ιουνίου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη στιγμή, 1η Ιουλίου, και συμφωνήσαμε ότι Θέλουμε να λάβουμε αυτές τις εκθέσεις και να τις αναλάβει κάποιος εισηγητής. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος, η κυρία Τσέσκοβα είναι εδώ. Όντως, ε, η έκθεση Ντελάγκη δεν μας απασχόλησε πολύ, γι' αυτό και είμαστε πολύ μπροστά στο χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα όμω να σα πω ότι μπορούμε να καθυστερήσουμε ακόμα δύο μήνε τη συνάντηση των συντονιστών. όμω είπαμε ότι καλό θα ήταν να λυθεί η απόφαση. Οι εκθέσει θα πρέπει να κατανεμηθούν. Η πρόεδρη, η των πρόεδρων ενδεχομένως θα μας δώσει ακόμα δύο μήνες. Αλλά πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση Τσέσκοβα αύριο. Εγώ αυτό προτείνω. Καλό θα ήταν λοιπόν να συζητήσουμε τώρα. Αλλιώς δεν ξέρω πότε θα μας δοθεί το πράσινο φως για πιθανή αναβολή. Δίνω το λόγο στην εισηγήτρια για να μας μιλήσει για το σχέδιο έκθεσης. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις εξηγήσεις σας. Ήταν πάρα πολύ σημαντικές αυτές για μένα. Και είναι σημαντική αυτή η πληροφορία, διότι η έκθεση είναι έτοιμη Έγινε και σχετική ακρόαση στις 22 Απριλίου για το θέμα αυτό και κατά την άποψή μου ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Υπήρχαν ε, πολλές πολύτιμες πληροφορίες, τις οποίες θα πρέπει να αναλύσουμε περαιτέρω, οι οποίες προέκυψαν σε συνέπεια αυτές τις ακρόασεις. Και γι' αυτό ακριβώς ε, ανησυχώ που είμαστε έτοιμοι να ψηφίσουμε για την έκθεση αύριο, χωρίς ε, να δώσουμε στους συναδέλφους το περιθέριο να υποβάλουν τροπολογίες. Και Λυπάμαι γι' αυτό. Σαφώς και μπορώ να δεχτώ τη διαδικασία που προτείνετε κύριε Πρόεδρε, δηλαδή να γίνει συζήτηση για το θέμα σήμερα και να ψηφίσουμε ε, αύριο, αλλά πραγματικά θεωρώ ότι είναι κρίμα να υποχρεωθούμε, να πιεστούμε, να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία ε, αν όμως εσείς θεωρείτε ότι πρέπει να το συζητήσουμε σήμερα, ας το συζητήσουμε και ας ελπίσουμε να δείξουν αρκετή ανοχή οι συνάδελφοι και να ψηφίσουν την έκθεση χωρίς να τους δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν τροπολογίες. Θα μπορούν να υποβάλουν βέβαια τροπολογίες, αλλά μόνο πριν από την Ολομέλεια ε, του Ιουλίου οπότε και θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια. Πραγματικά όμως λυπάμαι που συνέβη κάτι τέτοιο, διότι το αρχικό χρονοδιάγραμμα για την έκθεση ήταν σαφές και υπήρχε και μία σαφής προθεσμία για τροπολογίες ε, και έτσι μπορούσαν οι συνάδελφοι κάλλιστα να υποβάλουν τις τροπολογίες τους. Θα ήθελα τώρα να πω κάτι για την έκθεση, η οποία είναι αρκετά εκτεταμένη. Στις 22 Απριλίου που έγινε η ακρόαση, Ακούσαμε αρκετέ νέε προτάσει και ιδέε και πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω όλου του συναδέλφου ε, που συμμετείχαν στην ακρόαση η έκθεσή μου κάνει μια απόπειρα να είναι πλήρης και γι' αυτό ακριβώς και την έχω ε, κατανείμει σε διάφορα κεφάλαια. Δεν θα σας τα διαβάσω φυσικά ένα προς ένα, διότι είμαι βέβαιη ότι είχατε τη δυνατότητα να δείτε την έκθεση στη γλώσσα σας. Για το πρόγραμμα δράσης Το βασικό ερώτημα είναι γιατί δεν έλαβε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μία θετική δήλωση αξιοπιστίας ε, το 2006. Αυτό είναι αποτυχία του σχεδίου δράσης, ε, μήπως δεν διαμορφώθηκε καταλόγος ε, ή δεν εφαρμόστηκε καταλόγος. Και τι, και τι είναι αυτό το οποίο θέλει να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Η Επιτροπή απάντησε στην ερώτησή μου Και γνωρίζουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το σχέδιο δράσης ολοκληρώθηκε το 2009 και τρία από τα προηγούμενα 16 προγράμματα δράσης δεν μπόρεσαν να εφαρμοστούν, αλλά εφαρμόστηκαν με άλλο τρόπο. Κοινέ ε, αρχές εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες ετοιμάστηκαν και συμπεριλάφθηκαν στον αναθεωρημένο δημοσιονομικό κανονισμό. Αντίστοιχα, ασχολήθηκαν και με τα θέματα των ε, ε, δηλώσεων αξιοπιστίας εθνικής ε, διαχείρισης. Το όλο σχέδιο δράσης όμως θα πρέπει να το εξετάσουμε από τη σκοπιά της μείωσης των σφαλμάτων και εδώ δεν έχει γίνει δυστυχώς κάτι θετικό διότι η συχνότητα των σφαλμάτων αυξάνεται. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι θα προτιμούσε να υπάρξει μια θετική δήλωση αξιοπιστίας και φυσικά αυτή είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καθορίσει και ποιε είναι οι προποθέσει προκειμένου να λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θετική δήλωση αξιοπιστία και νομίζω ότι ήταν αρκετά ρεαλιστής στου στόχους του. Θα πρέπει όμως να αναλύσουμε την προσέγγιση του. Θεωρώ ότι η ουσία των όσων πρέπει να γίνουν είναι ε, να απλουστευθούν κάποια πράγματα. Στην έκθεσή μου ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόζει το άρθρο 32 του Δημοσιονομικού Κανονισμού πλήρως, διότι αυτό θεωρώ ότι θα βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εντοπίσει ποιες είναι δυναμίες στα συστήματα ελέγχου των κρατών μελών και από εκεί και πέρα να προτείνει περαιτέρω διορθωτικές ε, δράσεις για τους ολοκληρωμένους εσωτερικούς ελέγχους. Ε, καλό επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απλουστεύσει τις διαδικασίες στα αρμόδια τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να ε, προσπαθήσει να είναι πιο συγκεκριμένη όταν καθορίζει ποιο είναι το έργο των εθνικών ελεγκτικών αρχηχών. Έγινε μια συζήτηση εδώ τον Απρίλιο στη διάρκεια της ακρόασης και από τη συζήτηση αυτή προέκυψε και το θέμα της συνέχειας της διαδικασίας απαλλαγής του 2011. Θεωρώ ότι υπάρχει δυνατότητα πρόοδου στο μέλλον. Θεωρώ ότι ε, η έκθεση ε, για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ε, για τη δήλωση αξιοπιστίας θα πρέπει να ε, προετοιμαστεί εγκαίρως ώστε να μπορέσει να την αναλύσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία στόχο έχουν τη μείωση του ποσοστού σφαλμάτων. Η Ευρωπαϊκή όμως Επιτροπή μας είπε ότι Συγγνώμη, το ελεγκτικό συνέδριο είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να ε, εξετάσουμε ε, τα σφάλματα αυτά καθ' αυτά αν δεν έχουμε δείκτες ε, αξιοπιστίες. Γι' αυτό λοιπόν και ζήτησα να συσταθεί μια ομάδα εργασίας που θα περιλαμβάνει εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για να μπορέσουν να εγκρίνουν μέτρα ώστε να μπορέσουμε να έχουμε ένα προϋπολογισμό που θα βασίζεται στους δείκτες επιδόσεων. Βέβαια, ο ευρωπαϊκό ε, προπολογισμό που θα βασίζεται σε δείκτε επιδόσεων είναι ένα μακροπρόθεσμο στόχο. Θεωρώ σαφώ ότι πρέπει να συνεργαστούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό είναι προφανέ άλλωστε, αλλά η διαδικασία κατά την άποψή μου θα πρέπει να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι κοινό σχέδιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το υγιή μέλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει πάρα αυτά τι εργασίε τη. είτε με τροποποίηση στις συνθήκες είτε χωρίς τροποποίηση. Και κάποιες άλλες παρατηρήσεις τώρα. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή θα πρέπει να βοηθήσει ώστε να αλλάξει η νοοτροπία. Αυτό προσπαθώ να εξηγήσω και στην αιτιολογική μου έκθεση. Διότι είναι σαφές ότι το σύστημα το οποίο είναι ενισχύει αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτό το έχουμε πει επανειλημμένος, το έχουμε πει και κατά τη διάρκεια της ακρόασης εδώ τον Απρίλιο και είναι προφανές ότι πρέπει να αναζητήσουμε άλλες διαφορετικές αξίες σε αυτό το πλαίσιο. Και θα ήθελα επίσης να σας παραπέμψω στο άρθρο 21 της εκθεσής μου, Αναφέρεται μια δήλωση εκπροσώπου του ελεγκτικού συνεδρίου και στο σημείο 25 αναφέρομαι στην ε, μέτρηση της απόδοσης. Αυτές είναι οι ιδέες οι οποίες προέκυψαν από ένα μήνα εδώ στην ε, ακρόαση. Κατά την άποψή μου είναι καινοτόμα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε περαιτέρω. Σαφώς βέβαια θα πρέπει να υπάρξει και συνένεση προκειμένου να ε, εγκριθούν αυτές οι ιδέες και φυσικά αυτό δεν θα γίνει μια ανοιχτή. Θεωρώ όμως ότι το 2% το όριο του 2% για όλες τις πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό είναι ένα ε, ποσοστό το οποίο δεν αποφέρει αποτελέσματα και αυτό γιατί οι εθνικές ελεγκτικές αρχές ε, ουσιαστικά μειώνουν τεχνικά, τεχνητά το ποσοστό σφάλματος. Επομένως, θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλες προσεγγίσεις οι οποίες εξαρτώνται από την ε, ε, πολιτική κάθε φορά. Τουλάχιστον εγώ κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα μετά από τις απόψεις των εμπειρογνωμόνων που άκουσα στη διάρκεια της ακρόασης ε, του Απριλίου. Ευχαρίστως λοιπόν και εδώ να ευχαριστήσω και εκ των προτέρων τους συναδέλφους Θα προσπαθήσω να δείξω υπομονή. Ε, τι εννοώ, θα συζητήσουμε το θέμα σήμερα και πρέπει αύριο το πρωί να το ψηφίσουμε. Ελπίζω οι συνάδελφοι να συνειδητοποιούν ότι δεν φταίω εγώ. Ε, το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν τελείως διαφορετικό και η έκθεση αυτή είναι πολύ διεξοδική και εγώ δεν θα είχα επιτρέψει να συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή να μην δώσω τη δυνατότητα στους συναδέλφους να καταθέσουν ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ και ευχαριστώ για την υπομονή και την κατανόησή σας. Ναι. Ποιος θέλει το λόγο, Ζων Γιάννης Σκάιρ. Χαίρομαι. Συζητούμε αυτή την έκθεση γιατί ξεκινάει μια χρήσιμη, απαραίτητη συζήτηση που ξεκινήσαμε με την αχρώση. Πρόκειται για τις δηλώσεις αυτές και το θέμα είναι πώς μπορούμε να καλύψουμε κάποια κενά. Είδαμε από την ακρόση ότι όσον αφορά τη δήλωση αξιοπιστίας πολλές φορές κάποια ηχεία έχουν τεθεί αφαίρετα, παραδείγματο χάρη αυτό το 2% στο οποίο αναφέρθηκε και η συγκήτρια. Και βεβαίως εδώ ο καθορισμός αυτού του ποσοστού δεν ξέρω αν έχει γίνει βάση κριτηρίων ε, ή είναι κάτι που μπορούμε να το αμφισβητήσουμε και να το συζητήσουμε. Τώρα, πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας Αναφέρθηκε η συγγετρία σε κάποιες ανησυχίες. Ναι, μπορούμε να υποβάλουμε τροπολογίες και στην Ολομέλεια και αν προετοιμαστεί σωστά ο κατάλογος ψηφοφορίας μπορούμε να αποφύγουμε να πάμε προς μια κατεύθυνση που δεν είναι επιθυμητή. Πιστεύω ότι θα πρέπει εδώ να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Αν κατάλαβα καλά, αυτό θέλει και η συγκήτρια. Είναι πολύ σύντομη, αν θέλετε, η ο χρόνος που έχουμε και πραγματικά δεν ξέρω, συζητάμε σήμερα, ψηφίζουμε αύριο, αν θα προλάβουμε να υποβάλουμε και τις τροπολογίες όταν πρέπει. Ο κύριος Σοντή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Οι πρώτες μου κουβέντες για να ευχαριστώ την κυρία Τσέσκοβα και για το ενδιαφέρον που δείχνει σε όλα αυτά τα θέματα, τα περίπλοκα. Θα ήθελα να συμφωνήσω στα όσο είπε ο κ. Γκάιερ για τις προθεσμίες, γιατί είναι σπάνιο να αφαιρείται το δικαίωμα για υποβολή τροπολογιών από τους βουλευτές. Δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Εν πάση περιπτώσει, άλλε προτάσει μπορεί να υπάρχουν. Μια κρατή επιτροπή, παραδείγματι, μια ειδική επιτροπή. Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού θα μπορούσε να κάνει μια έκτακτη συνεδρίαση ένα Στρασβούργο τη Δευτέρα ή κάτι τέτοιο για να μπορέσουν ε, να έχουν το περιθώριο να τοποθετηθούν οι βουλευτές. Και τρεις παρατηρήσεις. Ωστόσο ότι πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειες μας για την αποδοτικότητα. Το είδαμε και με τις ακροάσεις. Είπαμε ότι θα επικεντρωθούμε στην ε, αποδοτικότητα, στις επιδόσεις και θα μας βοηθήσει και στην απαλλαγή. Εγώ είμαι επιφυλακτικό όπω προσέγγιση αυτή, γιατί το να έχει κανεί καλέ επιδόσει δεν σημαίνει απαραίτητα ότι οι αιτήσιοι λογαριασμοί ή οι δραστηριότητες που αυτοί εκφράζουν είναι εντάξει. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι καλέ επιδόσει επειδή είναι καλοί οι λογαριασμοί, ούτε ότι είναι κακέ όταν οι λογαριασμοί δεν είναι ικανοποιητικοί. Δεν υπάρχει άμεση ε, αιτιότητα. Έχω δει εγώ από την προσωπική μου ε, δραστηριότητα, την επαγγελματική μου δραστηριότητα και την εμπειρία ότι υπάρχουν τους πολύ καλοί λογαριασμοί, αλλά οι δραστηριότητες να είναι τελείως ε, λάθος. Και έτσι, και καθώς θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση της λειτουργίας, άλλωστε το είναι υποχρεωτική αυτή λόγω της συνθήκης, θα πρέπει να λύσουμε στο θέμα αυτό. Ε, δεν έχω σε αυτό καμία επιφύλαξη, αλλά θα πρέπει να δούμε πάλι τη σχέση αιτία και αιτία του. Και επίσης τη σχέση με τις εθνικές αρχές που αναφέρονται στην έκθεση. Εγώ δεν ε, πιστεύω ε, ότι είναι χρήσιμες οι, δια, οι διακηρύξεις εθνικής διαχείρισης. Ε, τουλάχιστον δεν πρέπει να περιμένουμε ότι θα μας φέρουν πολλά. Το να πιστεύει δηλαδή κανείς ότι μια δήλωση, μια διακήρυξη εθνικής διαχείρισης θα βελτιώσει την ποιότητα της αλυσίδας του νοσογνωμικού ελέγχου που εν τέλει θα καταλήξει σε μια θετική ε, δήλωση εξοπιστίας δεν είναι πιστικό επιχείρημα για μένα. Χρόνια τώρα άλλωστε το ζητάμε και δεν βλέπουμε αποτέλεσμα. Για ρωτήστε και το ελεγκτικό συνέδριο τι φρονεί επί του πρακτέου, γιατί εάν ένας υπουργός υπογράψει μία δήλωση εθνικής διαχείρισης, τι είδους αξία έχει ως προς το δημοσιονομικό έλεγχο. Δεν είναι ανεξάρτητος υπουργός, δεν είναι εξάρτητο όργανο. Επομένως, τι είδους αξία μπορεί να έχει τέτοια δήλωση. Από την άλλη, λυπούμε, και ίσως αυτό θα ήταν καλό να το συζητήσουμε με τους φίλους από τα Εθνικά Κοινοβούλια, να λυπούμε λοιπόν που δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί μία σχέση ε, μια αναφορά από τα εθνικά ε, ελεγκτικά συνέδρια, γιατί εκεί έχουμε ένα παράγοντα δημοσιονομικού ελέγχου, όταν έχουμε τις σχετικές παρατηρήσεις των ελεγκτικών συνέδριων των εθνικών. Και κάτι άλλο. το ποσοστό σφάλματος, ανεκτό ή μη και τα λοιπά που έχουμε συστήσει επί πολλά συναπτά έτη. Οφείλω να ομολογήσω ότι με προβληματίζει η μέθοδος που ακολουθεί το συνέδριο. Λέτε ότι υπάρχει αρνητική δήλωση αξιοπιστία. Τι να σας πω, δεν νομίζω ότι προκύπτει αυτό ξεκάθαρα από την έκθεση. Ε, υπάρχει μια θετική αξιολόγηση στην αξιοπιστία των ε, λογαριασμών και γνωμοδότηση πιστετική ως προς την ομιμότητα των ε, εσόδων και μία γνωμοδότηση αρνητική ως προς τα δαπάνες. Αλλά σαν τελική δήλωση, συνολική δηλαδή, δεν βλέπω ότι μπορεί να προκύψει. Για τους λογαριασμούς αναφέρεται σε μια σημαντική πτυχή το ελεκτικό συνέδριο, για δε τις δαπάνες αναφέρεται στην έννοια του ποσοστού σφάλματος. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να επεξεργαστούμε μια γενική αξιολόγηση από την γνωμοδότηση του ορίου σφάλματος ή ανεκτού σφάλματος και της αξιολόγησης για να δούμε αν πράγματι είναι θετική ή όχι η αξιολόγηση. Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έκθεση της, τη συγχαίρω την εισηγήτρια και εκφράζω τη λύπη μου για το ότι μας η δυνατότητα για κατάθεση τροπολογιών. Ίσως, Πρόεδρε, εσείς και έχω κάθε εμπιστοσύνη στο πρόσωπό σας, να μπορέσετε να βρείτε μια λύση. Ίσως αν ψηφίσουμε αύριο μπορέσουμε να δούμε ε, τροπολογίες της Επιτροπής που θα έχουμε τη δυνατότητα να ψηφίσουμε κατευθείαν στην Ολομέλεια. Άλλη λύση δεν έχω να προτείνω. Κύριο Μίλντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ την συγγετρία. Αρκετέ οι παρατηρήσει μου είναι ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις της συγγετρίας. Κάποια θέματα όμω δεν αλλάζουν. είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει η δήλωση αξιοπιστίας και είναι αρκετή αυτή που λένε ότι δεν είναι χρήσιμο, η συνθήκη ορίζει ότι πρέπει να καταρτίζεται και όποιος δεν το θέλει θα πρέπει να φροντίσει να αλλάξει συνθήκη. Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Έτσι πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος. Και πάντως δεν έχω βρει συγκεκριμένη απάντηση. Φαντάζομαι ότι ε, εφαρμόζεται η αυτή μεθοδολογία με αυτή του ευρωπαϊκού προπολογισμού και στα κράτη-μέλη. Αν το υποθέσουμε λοιπόν αυτό, τι είδου θετική δήλωση αξιοπιστία μπορεί να περιμένουν τα κράτη-μέλη. Πόσα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να λάβουν θετική δήλωση αξιοπιστία. Υπάρχει κανεί εδώ από την Επίτροπη που θα μπορούσε να πει ένα ναι. Και για το θέμα του 2%. Βεβαίω υπάρχουν εύστοχα επιχειρήματα, εύλογα επιχειρήματα. που απαντούν ότι αυτό εξαρτάται από το θέμα κάθε φορά. Όταν έχουμε παραδείγματι μικρό συμβάσεις, πολυάριθμους όπως συμβαίνει με την ε, έρευνα και τη δυνατότητα ενός τελικού αποτελέσματος μέχρι το 2% μπορεί αυτό να φαίνεται λογικό. Και όπως και να έχει σε διεθνές επίπεδο αποδεκτό ποσοστό σφάλματος με το 2%. Άρα νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι καλό είναι να μην αποκλίνουμε. Να μείνει αυτό και να μην ε, το τροποποιήσουμε, απλώς να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Και παρακαλώ να μου δοθεί απάντηση ε, πόσες χώρες θα μπορούσαν να λάβουν θετική δήλωση αξιοπιστίας. Και αν δεν μπορεί να απαντήσει η Επιτροπή, ας απαντήσει το Συμβούλιο. Ο Πρόεδρος. Εκ μέρους Επιτροπής θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να σας παρακαλέσω κύριε Ραφ να λάβετε το λόγο. Παρακαλώ. Πρόεδρε ευχαριστώ κύριο Σκράφ. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κυρία Τσίσκοβα για την εξαιρετική έκθεση και ιδιαίτερα για την υποστήριξη προς την Ευρωπαϊκή για τη διαδικασία της απλοποίησης ήταν σαφέ νομίζω από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι υπάρχουν κίνδυνοι, ότι δεν μπορεί να γίνει απλούστευση στο νέο στο νομικό πλαίσιο, γιατί είναι πολλές οι τροπολογίε που δεν βοηθούν στη διαδικασία αυτή. Επίσης, ε, υποστηρίζουμε ιδιαίτερα αυτήν την ιδέα για μια νέα ε, νοοτροπία μεταρρυθμίσεων. Συνεργαζόμαστε και με το Κοινοβούλιο και με το Συμβούλιο για να βελτιώσουμε ιδιαίτερα την έκθεση του άρθρου 318 και επίσης ε, η κατάρτιση προϋπολογισμού, ή εγγραφή στον προϋπολογισμό, καλύτερα ανάλογα με τις επιδόσεις, είναι μια ιδέα πάρα πολύ χρήσιμη την οποία θέλουμε να προωθήσουμε. Επίσης Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα μας φαίνεται η ανακοίνωση για τις ικανότητες του συστήματος που θα εμφανιστεί το Σεπτέμβριο και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στο ποσοστό 2% και την ερώτηση του κυρίου Μίλντερ. Εάν λοιπόν εφαρμοζόταν τέτοια μεθοδολογία στα κράτη-μέλη και υπήρχε τέτοιου είδους ποσοστό 2% πόσες χώρες θα μπορούσαν να λάβουν θετική δήλωση αξιοπιστίας. Η παθητική ερώτησή σας κύριε Μιλντερ. Διότι δεν προβλέπουν κανονισμοί ή και συντάγματα τέτοιου είδου ε, ε, υποχρέωση σε κράτη-μέλη. Αλλά υπάρχει από το Ηνωμένο Βασίλειο η πιθανότητα ε, για τον Γενικό Λογιστή του Κράτους να απορρίψει τη δήλωση αξιοπιστίας στην αντίστοιχη για το ε, σύστημα ε, κοινωνική ασφάλισης εφόσον έχει ποσοστό άνω του του 100, του 2%. Επίσης, πολλά από τα κράτη-μέλη βλέπουμε ότι ακόμα και το 2% με δυσκολία το φτάνουν. Καλωσορίζει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την υποστήριξη που εκφράζει το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή σας για την υλοποίηση των νέων προδιαγραφών προϋποθέσεων στον δημοσιονομικό κανονισμό που ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν παραμένει, παραμένει σταθερά υψηλό το ποσοστό, να δώσουμε κάποιες μεθόδους ανάλυση για το τι μπορεί να γίνει και να βελτιωθεί η κατάσταση, του κόστου τι είδους ωφέλη, πλεονεκτήματα και τι μέτρα θα πρέπει να εισαχθούν προκειμένου να δοθεί λύση σε υφιστάμενα προβλήματα. Διμερός τώρα. Υποβάλαμε στην εισηγήτρια κάποια τεχνικά ζητήματα. Δεν θα αναφερθώ διεξοδικά σε αυτά. Απλώς θα ήθελα να επικεντρωθώ σε κάποια σημαντικά ζητήματα που πρέπει πιστεύω να ληφθούν υπόψη στην έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή για μας να μην δοθεί το μήνυμα ότι δεν φέρνει αποτέλεσμα. Η μεμονωμένη επαλήθευση των λογαριασμών. Θέλω να περάσω το πείγμα ότι δεν φέρνει ακόμη αποτέλεσμα. Δηλαδή πρέπει να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτόν. αλλά και με εισαγωγή των απαραίτητων βελτιώσεων. Γι' αυτό λοιπόν το ακόμη στο σημείο 10 της εκθέσεως θα παρακαλούσα να ενσωματωθεί. Και επίσης το ότι τα συστήματα των κρατών μελών ε, τώρα δεν λειτουργούν στο πλήρες δυναμικό τους. Την ίδια παρατήρησα την είχα και για το σημείο 13, επίση Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι δεν υπάρχει ουσιώδης απόκληση μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς το, την εφαρμογή προληπτικών αφενός ή διορθωτικών αφετέρου συστήματος και εμείς από την Επιτροπή θέλουμε να προλάβουμε τα σφάλματα. Εάν λοιπόν, λοιπόν ένδειξη ουσιώδους απόκλησης μπορεί με την ετήσια διαδικασία ε, το ελεκτικό συνέδριο εφαρμόζει μια, μια αιτήσια διαδικασία με βάση συνθήκη, ενώ η Επιτροπή την πολυετική προσέγγιση. Όπως και να έχει, έχουμε αποστείλει τις παρατηρήσεις μας στην εισηγήτρια και στη γραμματεία της Επιτροπής σας και θα θέλαμε να αναπτύξουμε το διάλογο για να συζητήσουμε το πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη στη δικασία αυτή. Επίσης συστήθηκε το κατά πόσο είναι δυνατόν να δοθεί μια θετική δήλωση αξιοπιστίας. Εδώ θα παραπέμψω στη δήλωση που ακούστηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και στην οποία κάνατε εξής την αναφορά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ για τις ε, διευκρινήσεις του κ. Γκράφ για το σημείο 10 της εκθέσεως. Δεν καταγράφει νομίζω πιστά αυτά τα οποία είδε το ελληνικό συνέδριο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχαν ε, καταθέσει στην ε, ε, ακρόαση. Βλέπω να εμφανίζονται ξαφνικά φάσματα του παρελθόντος που δεν είχαν θέση εδώ. Με το θέμα του single audit. Εάν λοιπόν μείνει έτσι το σημείο 10, φοβούμαι ότι θα περάσουν πολλά χρόνια πριν ξαναδιορθώσουμε την πορεία μας. Θα έχουμε μπει σε τελείως λάθος τρόμο. Ελπίζω να μην συμβεί αυτό. Το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσουμε από εδώ και μπρος. Η Επιτροπή με την ανακοινήσή της για το single audit ήταν ε, πρώτη φορά η πρόταση το 2004 και το ερώτημα είναι πώς συνεχίζουμε με αυτή την παλαιά ιδέα και έννοια Μα είπατε ότι δεν φτάσαμε ακόμη. Ναι, ευχαριστώ πολύ για τη διευκρίνηση. Νομίζω ότι τα είχαμε καταφέρει. Ερωτώ λοιπόν πώ θα τα καταφέρουμε, πώς θα περάσει και πώς μπορούμε να πείσουμε και τα κράτη-μέλη για να βελτιωθεί και το σύστημα των κυρώσεων αλλά και των ελέγχων. Πώς ή τι πρέπει να αλλάξει προκειμένου να αλλάξουν τα κράτη-μέλη νοοτροπία αλλά πάνω απ' όλα και οι αρχές τους για να φέρει αποτέλεσμα τελικά αυτή τη προσπάθεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιο άλλο το λόγο. Τότε θα παρακαλώ τον κύριο Γκράφνα αλλά αυτό το λόγο να απαντήσει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά την ερώτηση αν θέλει ακόμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόσει τις ιδέες του Single η απάντηση είναι σαφέστατα ναι. Αν ε, αναλύσουμε το σχέδιο κανονισμών που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δηλώνεται σαφώς ότι πρέπει να βασιστούμε στο έργο των ελεγκτικών αρχών ε, σε θέματα συνοχής ε, και στους οργανισμούς πιστοποίησης στη Γεωργία. Αν δείτε και την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκεί διαφαίνεται σαφώς ότι μπορούμε να βασιστούμε στο 70% ε, των εγγράφων ε, των ε, γνωμοδοτήσεων από τους ελέγχους που γίνονται. Αν τα διαβέστε ανάποδα, το 70% των στατιστικών στοιχείων σφάλματος που παρουσιάζονται από τα κράτη-μέλη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρηθεί τα στοιχεία βάσει των αποτελεσμάτων ε, της δικής της της δουλειάς, ε, των αποτελεσμάτων του ελεγκτικού συνεδρίου και από εκεί παράγονται νέα στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι πολύ εγκύτερα στα στοιχεία που μας δίνει το ελεγκτικό συνέδριο ε, και το ποσοστό σφάλματος δηλαδή είναι πολύ ψηλότερο. Τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να μας δίνουν πιο αξιόπιστες πληροφορίες. Εδώ πρέπει να πούμε ότι δραστηριοποιείται έντονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείνει ε, δημοσιονομικές διορθώσεις. Αν δείτε για παράδειγμα τους λογαριασμούς για το 2013, ε, διαπιστώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βάλει δημοσιονομικές διορθώσεις που ανέρχονται στο ποσό των 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Εάν λοιπόν τα κράτη-μέλη δεν ε, διασφαλίσουν ότι έχουν υγιή συστήματα, ε, τους επιβάλλονται κυρώσεις ε, μέσω δημοσιονομικών διορθώσεων και φυσικά αυτά τα ποσά δεν είναι καθόλου ασήμαντα, είναι ίσα ίσα πολύ σημαντικά ποσά. Στην παράγραφο 10, στην παράγραφο 10 ε, και 13 ε, γίνονται οι αλλαγές αυτές. Ελπίζω να ήμουν αρκετά σαφής και να διαπιστώσετε τι σκοπεύει να κάνει η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή στο μέλλον για να εφαρμόσει και το single audit. Ευχαριστώ. Δεν τα κάποιο άλλο το λόγο. Νομίζω. ότι το βασικό καθήκον μας είναι να φτάσει αυτή η έκθεση στην Ολομέλη αυτή τη στιγμή αλλά είναι κοινή προσπάθεια της Επιτροπής μας. Θέλουμε όλοι να συζητηθεί αυτό το θέμα και ελπίζω να μπορέσουμε να έχουμε τροπολογίες στην Ολομέλεια. Να δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια αν θέλει να σχολιάσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Δύο-τρία σχόλια στα όσα ακούστηκαν. Καταρχάς, Πραγματικά θα ήθελα να στηρίξει την έκθεση η Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια. Κάποιος συνάδελφος αναφέρθηκε στη δήλωση αξιοπιστίας. Αν θεωρούμε ότι είναι ένα λογικό εργαλείο ή όχι. Ή αν αυτό το όριο του 2% Κοιτάξτε, θα μπορούσε κάλλιστα να πει κάποιος ότι θα μπορούσε να είναι το ποσοστό σφάλματος, το όριο σφάλματος 2,5-3%. Είναι κάτι το οποίο συζητήσαμε και στην ακρόαση και νομίζω ότι είναι μια συζήτηση η οποία πρέπει να μείνει ακόμα ανοιχτή. Ίσως να μην είναι δυνατόν ε, να βρίσκονται σε αυτό το όριο σφάλματος όλες οι ε, πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. και αυτό φυσικά μπορεί να οδηγήσει τα κράτη-μέλη να ε, μην χρησιμοποιούν το ποσοστό σφάλματος. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και για την πρότασή σας να συνεδριάσουμε πριν από την Ολομέλεια, αν δεν μπορέσουμε να συζητήσουμε τις τροπολογίες εδώ. Πραγματικά θα ήθελα να στηρίξω οποιαδήποτε πρωτοβουλία, οποιασδήποτε πολιτικής ομάδας ε, για να συνεδριάσουμε και πριν από την Ολομέλεια ε, για να συζητήσουμε τι τροπολογίε. Θα ήθελα να σα ευχαριστήσω όλους ε, για την εξαιρετική αυτή ιδέα. Αναφερθήκαμε επίσης και στο ε, στοιχεία των επιδόσεων. Είναι κάτι το οποίο είναι νέο στοιχείο στις εκθέσεις. Στο παρελθόν ασχολήθηκα αρκετά χρόνια με λογιστικά ζητήματα και ελέγχους και η προσέγγιση των επιδόσεων είναι μια προσέγγιση με την οποία δεν είμαι και τόσο εξοικειωμένη μεν, αλλά θεωρώ ότι έχει μέλλον δε. Η στάση που τηρούμε είναι μάλλον αυστηρή για το θέμα αυτό και βασίζεται σε τυπικά κριτήρια ε, και ε, θεωρούμε ότι βάσει αυτών δεν θα μας οδηγήσει στα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό όμως είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει στο μέλλον. Ε, το ακούσαμε και στην ακρόαση. Πρέπει να το συζητήσουμε περαιτέρω. Τώρα... Οι εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας είπε κάποιος ότι δεν είναι και τόσο σημαντικές εγώ νομίζω ότι θα πρέπει ε, τουλάχιστον ε, να αναγνωρίσουμε ότι έχουν μια πολιτική σημασία, ίσως όχι νομική σημασία ή ποινική σημασία, αλλά σε πολιτικό επίπεδο οι εθνικές δηλώσεις αξιοπιστίας θα πρέπει να έχουν κάποια βαρύτητα κατά την άποψή μου, διότι εάν ο Υπουργός Οικονομικών ε, είναι αυτός ο οποίος υπογράφει στη δήλωση αξιοπιστίας, ε, θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι έχει μια κάποια βαρύτητα. Τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για το 80% του προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα τις μεθόδους του ελεγκτικού συνοδρίου για τη δήλωση αξιοπιστίας, ε, νομίζω ότι αναφέρθηκα σε αυτό και προηγουμένως, στην προηγούμενη παρέμβασή μου. Δεν είναι αρκετά σαφές, ε, μπορούμε να το συζητήσουμε περαιτέρω. Το σχέδιο δράσης εγκρίθηκε πριν από αρκετά χρόνια και φαίνεται ότι δεν είναι πλέον ε, απόλυτα ρεαλιστικό. Ίσως θα ήταν πιο λογικό να ήταν διαφορετικές οι, προθέσεις, οι προϋποθέσεις ε, εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκράφτ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι αυτό το γετ το οποίο ανέφερε, αυτό το ακόμα, θα μπορούσε ίσως να συμπεριληφθεί στην έκθεσή μου. Στην ακρόαση όμως του Απριλίου ακούσαμε και κάποιους να ισχυρίζονται ότι ε, η μέθοδος του single audit κατά, κάποια, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχει αποτελέσματα. Θα εξακολουθήσει να είναι αρνητική η δήλωση αξιοπιστίας, ε, θα εμείνουμε σε αυτό το όριο σφάλματος του 2% και το single audit θα αποτύχει. Αυτά λοιπόν. Ευπρόσδεκτες όλες οι τροπολογίες που θα θέλετε να υποβάλλετε. και ίσως ε, η αρχή της, ε, των επιδόσεων ή οποιαδήποτε άλλη αρχή να μας οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Είναι δύσκολο να το προδικάσουμε αυτό από τώρα. Παρ' όλα αυτά θα ήμουν ιδιαίτερα ευτυχής αν μπορέσετε να προσθέσετε κι εσείς το οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό για την έκθεση αυτή. Διότι γνωρίζω ότι πολλά από τα μέλη της Επιτροπής έχουν ευρύτατες γνώσεις και πολλοί από εσάς βρίσκεστε εδώ πολύ περισσότερο καιρό από μένα. Και μία τελευταία ερώτηση προς την κυρία Γκρέσλε. Συμφωνώ ότι η ποιότητα των ελέγχων θα πρέπει να είναι καλή σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώντας από το βασικό επίπεδο στα κράτη-μέλη, περιφερειακό επίπεδο, τοπικό και από εκεί και πέρα ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Το ιδεώδες βέβαια θα ήταν να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για όλους αλλά αυτό μάλλον δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να επιτύχουμε προς το παρόν ή τουλάχιστον όχι στο εγγύς μέλλον. Συμφωνώ ότι το single audit όμως ε, το χρειαζόμαστε κατά πάσα πιθανότητα. Χρειαζόμαστε ένα ενίο πλαίσιο διότι ε, μας ενδιαφέρουν τελικώς τα ίδια ποσά. Σας ευχαριστώ όλους αγαπητοί συνάδελφοι. Και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν είχαμε περισσότερο χρόνο να συζητήσουμε το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια. Νομίζω τελειώσαμε και με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ πολύ όλους. Ήταν πολύ εντατική συνεδρίαση. Ευχαριστώ την ε, κυρία Τσέσκοβα για την έκθεση. Και πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η εντολή για τον τριμερή διάλογο. Πολύ σύντομα, λέει ο κύριος ε, Χάιερ. Ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν όλοι οι συνάδελφοι. Και νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε κάποια συμπεράσματα και να δώσουμε και κάποιες οδηγίες κατά κάποιο τρόπο στους συναδέλφους της Επιτροπής Προεπολογισμού όσον αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Θα πρέπει να συνεχίσουν να επεξεργάζονται τα σημεία που θα πρέπει να εξεταστούν περισσότερο, εκεί που υπάρχει κακή διαχείριση, εκεί που θα πρέπει να φτάσουμε σε κάποιες ε, καλύτερες ε, διαχειρίσεις. Το κείμενο μου συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα σημεία και νομίζω ότι το θέμα καλύπτεται ε, πλήρως. Ποιος θέλει να πάρει το λόγο, λέει ο Πρόεδρος. Δεν βλέπω κανέναν. Ο κύριος Σοντή. Δεν ξέρω αν αυτό το θέμα συμπεριλαμβάνεται εδώ, αλλά ένα σημείο που μας απασχολεί όσον αφορά το πλαίσιο μέχρι το 2020 είναι τα ποσά που εκκρεμούν από το 2013 και τα οποία θα επηρεάσουν το 2014. Μήπως πρέπει εδώ στην έκθεση αυτή να βάλουμε την παρατήρηση ότι για τον τριμερή διάλογο του 2014 θα πρέπει να συμφωνήσουμε όσον αφορά τα ποσά που λείπουν, τουλάχιστον στις επαφές μας με τις κυβερνήσεις. 13, 14 δισεκατομμύρια, ακόμα διάφορους αριθμούς. Εγώ πρότεινα στον Αλάνα Μασούρ, βάσει των υπολογισμών της Επιτροπής, θα πρέπει να έχουμε πιστοποιητικά δημοσιονομικού ελέγχου, να μας πούν πρόκειται για 13 ή για 14 δισεκατομμύρια. Ακούω υπουργού να λένε 8 ή 9 δις θα πληρώσουμε κάποια ποσά το 2013 και τα υπόλοιπα θα πια πραγματευτούμε για το 2014. Ξέρουμε όμως γιατί ποσό πρόκειται στο τέλος του 2013. Και τι θα μπει στο 2013, τι θα μπει στο 2014. Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού ίσως πρέπει εδώ τουλάχιστον να ελέγξει αυτό το ποσό που μας δίνει ο αρμόδιος επίτροπος. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε, αλλά έχω την εντύπωση ότι καλό θα ήταν να έχουμε ακριβώς την κατανομή των ποσών στο 13 και στο 14. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρέσλε. Η προθεσμία για τις τροπολογίες που είναι. Κοιτάξτε, δεν έχω θέμα. Για το, 7 σημείο, για το σημείο 7 θα έλεγα ότι είναι λίγο παράξενο. Εδώ βλέπουμε κράτη-μέλη που επιτέλους ε, υιοθετούν την αρχή της καλύτερης ε, χρήσης των κονδυλίων, better spending, και τους επικρίνουμε. Τι να πω, καταλαβαίνω τους σοσιαλιστές, αλλά εμείς εδώ σαν Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού τόσα χρόνια ζητάμε αυτή την καλύτερη διαχείριση, καλύτερη κατανομή και χρήση των κονδυλίων. Νομίζω λοιπόν ότι δεν πρέπει εδώ να υπονομεύσουμε οι ίδιοι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στην Ίνες. Ναι, να σχολιάσω αυτή την παρατήρηση για τους σοσιαλιστές. Δεν κατάλαβα προς τι αυτή η διευκρίνηση. Ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε μια σειρά από καταγγελίες που λάβαμε για την κακή χρήση των διαστατικών ταμείων της γερμανικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Να μην είναι μόνο οι σοσιαλιστές ε, αυτοί οι οποίοι θα μιλούν για την καλύτερη χρήση των ε, δημοσίων οικονομικών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γκάιερ, θέλετε και εσείς. Θα ήθελα όμως εγώ να αναφερθώ στις διαπραγματεύσεις και στο βαθμό ενημέρωση που έχουμε για την εξέλιξη στις διαπραγματεύσεις σε σχέση με τα όσα βλέπουμε και στα μέσα μας Τι μεταφέρεται στις ομάδες από τους βουλευτές. Έχεις εσύ κάποια ανάμειξη ως ε, αρμόδιος για την γνωμοδότηση. Εύκολα να απαντήσω στη τελευταία ερώτηση. Είμαι μέλος και της Επιτροπής των Προϋπολογισμών. Και εκεί οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές συνομικό πλαίσιο και τις, ε, τα, τα προβλήματα ως προς τον προϋπολογισμό του 2014 πάλι στο ίδιο θέμα έγκυνται. Είναι αλληλένδετα δηλαδή, όπως λέει το Κοινοβούλιο, προβάλλοντας την επιχειρηματολογία ότι οι μεγάλες διαφορές μεταξύ υποχρεώσεων και πληρωμών που παρουσιάζουν τα κράτη στα πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το διαρθρωτικό έλλειμμα είναι αυτό το οποίο θα δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα, έτσι νομίζω λέγει ο κύριος Οντζή. Στο παρελθόν είχαμε πάντοτε ταυτίσεις, τα ποσά των δεσμεύσεων υποχρεώσεων και των πληρωμών. Τώρα είναι σαν να λέμε ότι είμαστε διατεθειμένοι να αναθέσουμε έργα 960.000 δισεκατομμυρίων ευρώ, αλλά τα 908 μόνο δις θα μπορέσουν να πληρωθούν. Θα περισσεύουν δηλαδή, θα λείπουν καλύτερα 2 εκατομμύρια στην τελική πληρωμή. Και άρα όταν έρθει η ώρα να ολοκληρωθεί ένα έργο, υπάρχουν βέβαια και νομικέ δυσκολίε, καθυστερήσει και όλα αυτά τα πράγματα μπορούν να προκύψουν κάποια στιγμή. Μια απόκληση δηλαδή μεταξύ της ε, ε, υποχρέωσης και της ε, πληρωμής, αλλά το ερώτημα είναι μήπως πρέπει τελικά να ανησυχούμε για την νομιμότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ε, επιδίωξη των πολιτικών της στόχων. Το Κοινοβούλιο μπορεί να λέει, εν προκειμένου, ότι εφόσον τώρα, όπως έχει το πρόβλημα, με την ίδια αιτία, είμαι διατηθειμένο να προσπαθήσω να αντιμετωπίσω με το ίδιο σύστημα, δηλαδή τον διορθωτικό προπολογισμό, αμφισβητώ, ε, θέτω σε κίνδυνο την αξιοπιστία της ίδιας της Ένωσης. Πρόβλημα επίση είναι ω προ το εξή ότι εμεί βέβαια από την Επιτροπή προπολογισμών πάντα πιέζουμε με απειλέ την Επιτροπή και τον Επιτροπό Λεβαντόφσκι ως προς την παρουσίαση διαφορετικών αριθμητικών. Πρώτα ακούγονται 16 δις, μετά 15 κτλ. με αποτέλεσμα να καταλήγουμε στην υποψία ότι μάλλον τους αριθμούς δεν τους ορίζουν τα μαθηματικά αλλά η πολιτική. Και έτσι περιμένουμε να δούμε αν η Επιτροπή εν τέλει θα είναι σε θέση να καταβάλει το τίμημα, να πληρώσει τις πολιτικές εκείνες, να δηλώσει τη βούληση να πληρώνει τις πολιτικές που θέλουμε να υλοποιήσουμε και αντίστοιχα να ασκήσει την πίεση και στο Συμβούλιο, όπου εν τέλει και εμείς θα φαινόμασταν. Θα αποφεύγαμε μάλλον να φανούμε σαν τον ε, ε, σαν την Μωρή Παρθένο όταν τελικά η Επιτροπή θα έλεγε «Α, τι είχαμε πει 15, όχι, τελικά θέλαμε λιγότερα» κτλ. Και θα άρχισε μετά να τα κόβει φέτες για να δώσει πρώτα 7 και μετά ακόμα λίγα και λίγο περισσότερα γιατί υποτάσσεται σε κάποιες ε, βουλείς του Συμβουλίου. Έτσι λοιπόν είπαμε στο Λεβαντόφσκι και ξεκάθαρα τα εκφράσαμε την απειλή μας αν δεν μείνει στο ποσό που θα πεις να έχεις υπόψη θα έχει συνέπειε. Αυτό για να αποφύγουμε τις πολιτικές ε, υπαγορεύσεις στο θέμα αυτό. Βέβαια το έχουμε συζητήσει και με το Γενικό Διευθυντή και φαίνεται ότι συνεννοούμαστε. Καταλαβαίνω λοιπόν τα πολιτικά προβλήματα και επιφυλάξει του κύριου Οντή, αλλά... Είναι ένα θέμα αυτό το οποίο η Επιτροπή των Προϋπολογισμών ναι, μπορεί να βάλει μέσα στην έκθεσή της, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε περισσότερο χωρίς να έχουμε πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο και να πούμε ότι αφήνουμε περισσότερο, ότι παίρνουμε τη νομική βάση την οποία έχουμε με το 213 συμπληθωρισμό, του, με το 2013 συμπληθωρισμό και βλέπουμε μετά πώς θα προκύψουν ε, τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων. Αυτή η κατάσταση κινδυνεύει να μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Αλλά από την άλλη, ο καθένας πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Απαντήσεις ουσιαστικές δεν παίρνουμε. Και το να πιστέψουμε αυτά που λέγονται χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο μας φαίνεται υπερβολικό. Το έχω περιλάβει όλο σε από τα εκθεσέω μου. Αυτά. Προς το παρόν, βέβαια, αν κοιτάξουμε αυτοί που ζητούν να αξιοποιούνται καλύτερα τα κονδύλια, το τι ακριβώς θέλουν σαν τελικό στόχο, που είναι η περικοπή εν γέννη του προπολισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η περιστολή των δραστηριοτήτων της εν τότε διαρωτώ με τι προσπαθούν να κάνουν. Μέσα στο Συμβούλιο προσπαθούν να περικόψουν, κάνουν μια συζήτηση μεταξύ ομολόγων στο Συμβούλιο όπου συζητούν ποιο είναι το καλύτερο management και πότε γίνεται και πότε δεν γίνεται. Το ερωμένο Βασίλειο Φερρυπίν, το οποίο γανακτισμένο διατυπώνει τις αντιρρήσεις και τα σχόλιά του για το πόσο κακό, κακό διαχείριση υπάρχει στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, και μετά κάποια ποσά τεράστια, δεν πω νούμερο γιατί δεν θα κάνω λάθος σου, αλλά πολλά εκατοντάδες εκατομμύρια φαίνεται να έχουν χαθεί από τον Βρετανικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, μην προσπαθούμε τώρα να συζητούμε πράγματα περιτά. Ας κάνουν και αυτοί που θέλουν καλύτερη διαχείριση του ευρωπαϊκού χρήματος, από πλευράς τους το καθήκον τους, ας μην παρουσιάζουν την κατάσταση στο εσωτερικό τους ιδεώδη και ότι τάχ κάποια άλλα κράτη τους ζητούν συνέχεια να δίνουν λεφτά. Το better spending αυτό, friends of better spending, ε, εν χαρακτηρίζει μια συγκεκριμένη προσέγγιση και αξιολόγηση. Βεβαίως όλοι θέλουμε μια καλύτερη αξιοποίηση και απορρόφηση των κονδυλίων, αυτός είναι ο στόχος όλων μας. Σε αυτό πάνω εργαζόμαστε. Αλλά τουλάχιστον όσο όποιοι θέλουν στο Συμβούλιο να το επιδιώξουν αυτό, ας έχουν φροντίσει πρώτα στο εσωτερικό τους να βελτιώσουν την κατάσταση. Ο Γενικός ε, Διευθυντής της Περιφερειακής Πολιτικής μας είπε ότι από τα 18 από, ε, από τα κράτη-μέλη 18 δεν έχουν ε, καλή διαχείριση των περιφερειακών και από αυτά τρία ήταν Friends of Better Spending. Βρετανία, Γερμανία, 100 ε, τι άλλο να πω. Μάλιστα. Ωραίο, ωραίο black humor αυτό. Κυρία Γέγκλερ. Κυρία Γέγκλερ. Γκρέσλε. Ναι, ναι, ναι. Αν ήταν αυτό βέβαια το θέμα δεν θα είχα καμία αντίρρηση. Αλλά το να ξεκινήσουμε ένα νέο θέμα στο οποίο τίποτα δεν είναι δεδομένο, τι να σας πω. Θα ήθελα να επισημάνω λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο έχει δεχθεί ένα κενό, μια απόκληση 15 δις μεταξύ των υποχρεώσεων και των πληρωμών. Αυτό είναι πάγια τακτική, έχει συμβεί πολλές φορές και στο παρελθόν, μπορεί να γίνει δεκτό και στο «Όχι» λέει ο πρόεδρος, «Όχι δεν έχετε δίκαιο». Να σας πω, εγώ δεν το είχα δεχθεί αυτό το gap, αυτό το κενό. Υπάρχει απο... Δεν υπάρχει όχι, δεν υπάρχει καμία απόκληση, έχει γίνει πάντοτε έτσι. Να σας πω, όχι το έχουμε δεχθεί, λέει η κυρία Γκρέσλε. Και πρόβλημα δεν υπήρξε ποτέ. Γιατί? Διότι δεν έχουμε ποσοστό συγχρηματοδότησης. Δεν χρησιμοποίησαν δηλαδή τα, τα, τα κράτη το ποσό αυτό. Και θα ήθελα ένα τεχνικό πρόβλημα να το συζητήσουμε ως τεχνικό και όχι ως πολιτικό. Γιατί δεν είναι πολιτικό. Αυτό ήταν ο κύριος, η κύρια προσπάθεια σε ένα τεχνικό πρόβλημα να το χαρακτηρίσουμε πολιτικό και να μπλέξουμε τη συζήτηση ακόμη περισσότερο. Ας είμαστε λοιπόν πιο ε, στο ψητό στην ουσία και ας αφήνουμε τις περικοκλάδε. Και θα ήθελα να αναφέρω ότι το θέμα του λαθρεμπορίου προκαλούν οι ίδιες οι εταιρείες της καπνομηχανίας. Βεβαίως και θα πρέπει να μας απασχολήσει, βεβαίως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και βεβαίως θα πρέπει να δούμε αυτή η συμφωνία που έχει συναυθεί, γι' αυτό άλλωστε συνήφθη, με την καπνομηχανία, τι είδους αποτέλεσμα φέρνει. Εφόσον υλοποιείται σωστά, είναι πολύ θεμητό το ερώτημα. Από την άλλη βέβαια, μπορεί και το ελεγκτικό συνέδριο να μελετήσει πολύ προσεκτικά και ήρεμα τι είδους ε, δράσεις εκδηλώνουν αυτές οι επιχειρήσεις καπνιδομηχανίας πέραν της σχετικής συμφωνίας εάν εκτός από τη συμφωνία κάνουν και στο περιθώριο κάποιες άλλες δραστηριότητες λαθρεμπορίου. Για το better spending δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που είπατε, αλλά ε, εάν ε, οι επικρίσεις φυσικά είναι ίδιες με τις δικές μας, ας μην τις προσαρμόσουμε όλα με την ιδεολογία μας. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Έχω κι άλλες δύο ερωτήσεις. Οι πραγματικοί φίλοι όμως του Better Spendings είμαστε εμείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Γιάννης Γκάιερ έχει δίκιο όταν λέει ότι στο Συμβούλιο ακούμε διάφορες διευθετήσεις του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πώς ε, τα κονδύλια ιστρέων, πώς ε, τελικά πρέπει να δαπανηθούν. Θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά στον δικό μας τομέα αρμοδιότητας τι πρέπει να γίνει και τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, γιατί εδώ είμαστε για να προσπιστούμε τα κοινοτικά συμφέροντα. Και αν κοιτάξει κανείς παραδείγματος χάρη στη δική μας χώρα, που είναι μια ομοσπονδιακή χώρα, τα συμφέροντα των κρατηδίων και το γενικό συμφέρον, την εμπιστοσύνη και το γενικό συμφέρον της Ομοσπονδίας που πολλές φορές ε, αντικρούνται, που πολλές φορές δεν συμβαδίζουν. Εδώ, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να διασφαλίσουμε το γενικό συμφέρον, το κοινοτικό συμφέρον. Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να καθόμαστε εδώ. Αν πάψει να υπάρχει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε πραγματικά δεν έχει νόημα καμία περαιτέρω δράση. Ο κ. Μούλτερ και ο Ζαν Πιέροντι έχουν ζητήσει το λόγο. Πολύ σύντομα. Υπάρχει το σύστημα των δεσμεύσεων και των πληρωμών στο ευρωπαϊκό προπολογισμό. Όπως είπε ο Γιάννης, δεν μπορούμε να μην είμαστε συγκεκριμένοι όταν υπάρχει μια δέσμευση, θα πρέπει να υπάρχει η πρόβλεψη για την πληρωμή και η δυνατότητα πληρωμής. Οι αρμόδιες αρχές και τον προπολογισμό σήμερα γνωρίζουν μια περίεργη κατάσταση. Από τη στιγμή που εγκρίνει η αρμόδια αρχή του προπολογισμού μία δέσμευση, δεν μπορεί μετά να λέει δεν υπάρχουν τα κονδύλια για τις πληρωμές. Δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση στον κοινοτικό προπολογισμό. Και γι' αυτό και το νέο σύστημα για την διαχείριση των ίδιων πόρων είναι απαραίτητο κατά την άποψή μου. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Δεν υπάρχει αυτό το σύστημα, σας λέω. Δεν γίνεται να συνεχίσουμε έτσι. Ευχαριστώ πολύ, ο Ζων Ναι, πολύ σύντομο αναφορά αφορά τα, τις πιστώσεις δεσμεύσεων και πληρωμών. Υπήρχαν αυτά τα δύο συστήματα και όταν μιλάμε από πολιτικής απόψεως τουλάχιστον, μιλούσαμε για πιστώσεις δεσμεύσεων. Ο Βρετανός ουσιαστικά πρωθυπουργός είναι αυτός που άλλαξε την ορολογία και άλλαξε το σύστημα, γιατί έτσι γύρισε πίσω στη χώρα του και παρουσίασε χαμηλότερους αριθμούς. Εντάξει, αν συμφωνούμε όλοι, ας μιλούμε για τις πιστώσεις πληρωμών. Δεν χρειάζεται να υπάρξει εδώ διαμάχη για 3 ή 4 δισεκατομμύρια. Είναι τεχνικό το θέμα που συμφωνούν όλες οι χώρες για 7 δισεκατομμύρια. Τι κάνουμε με τη διαφορά. Τη γνωρίζω εγώ τη διαφορά. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έρευνας αποφασίσει να σταματήσει το προγραμματισμό, θα βρεθεί η λύση θα βρεθούν από εκεί τα κονδύλια. Αναρωτιέμαι λοιπόν μήπως ο εισηγητής δεν θα έπρεπε να βάλει μία αναφορά κάπου στην έκθεσή του πριν το τέλος του 2013 και το ξεκίνημα του 2014 να γίνει μία αξιολόγηση και να δούμε τι πρέπει να μπει σαν ποσό, τι παραμένει, 6, 7, 8 είναι το ποσό που θα βάλουμε για το 2013 το θέμα των πιστώσεων πληρωμών μέχρι το τέλος του 2013 πρέπει να ξεκαθαριστεί και πρέπει να υπάρχουν οι πόροι. Γιατί όταν λέμε ότι δεν θα μπορέσει να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μα αυτό είναι γελίο. Αν δεν μπορούμε να πληρώνουμε τα τιμολόγια, καταλαβαίνετε ότι έξι μήνες πριν τις εκλογές η αξιοπιστία μας έχει εξανεμιστεί. πολλά θέματα προς συζήτηση. Υπάρχουν τροπολογίες και θα ξεκινήσει η κανονική διαδικασία. Η Επιτροπή έχει κάτι καινούριο να μας πει. Έχετε κάτι το σοβαρό, το πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε. Αν όχι, τίποτα το καινούργιο δεν μπορώ να σας πω. Να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Οντή. Βεβαίω θα υπάρχει η έκθεση στο τέλος του χρόνου για την εκτέλεση του προϋπολογισμού και αυτό βεβαίως από το ελεγκτικό συνέδριο. Θα έχετε λοιπόν εκεί το ποσό που παραμένει και δεν έχει πληρωθεί στο τέλος του 2013. Ο κύριος Σοντή, να κοιτάξετε τώρα οι εκθέσεις του συνεδρίου Καταλαβαίνετε ότι αν φτάσουν το 2015 για το 2013 δεν θα είναι και πολύ χρήσιμο. Ωραία, λέει ο Πρόεδρος. Θα δώσω πάλι το λόγο στον εισηγητή. Όχι, δεν τον θέλει. Διακόπουμε λοιπόν και θα ξαναρχίσουμε αύριο το πρωί στις 9. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί στις 9 στην ίδια αίθουσα.